ο οποίος ε, μας εγκατέλειψε προχθές ε, το 1989 ήταν ε, αυτός που ξεκίνησε την Επανάσταση, κάτι το οποίο οδήγησε στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος και αυτό του έδωσε ένα κύρος ηθικό ιδιαίτερα μεγάλο. Ε, από παλιά είχε ξεκινήσει την κριτική προς την κομμουνιστική κυβέρνηση και το καθεστώς συχνά τον ε, επέκρινε αλλά και τον καταδίκαζε. Ήταν, αποτέλεσε πραγματικά ένα παράδειγμα και υπόδειγμα ανθρώπου σε ό,τι αφορά τον ανθρωπισμό του, τον, ε, την κουλτούρα του και πραγματικά επέκρινε έναν ε, άκρατο ηλισμό ο οποίος ε, επικρατούσε ανά τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να αποτίσουμε ενός λεπτού σιγή. Danke Προτού να περάσουμε στην μέσα διάταξη, να σας πω ότι έχουμε κάποιες τροποποίησεις. Ο κύριος ε, Λούντου δεν ε, θα μπορέσει να παραστεί και το ίδιο ισχύει για την γνωμοδότηση παντούς ε, για το θέμα που είχαμε στη μέσα διάταξη και θα θέλαμε να επιστρέψουμε και την αυριανή συνεδρίαση προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να επιστρέψουμε εγκαίρω στα σπίτια μας. Θα ήθελα λοιπόν όλοι να μπορέσετε να φύγετε χωρίς να χρειαστεί να εγκατρέψετε την αίθουσα άρων-άρων. Λοιπόν, μέχρι τις 4 και 4. Θα ακούσουμε την κυρία Ρέντινγκ. Μετά θα ακούσουμε την έκθεση της ε, Μάρκο, ε, συγγνώμη, της ε, κυρίας ε, Βερζιά, μετά την έκθεση Σκουρία. Να δώσουμε κατευθείαν τον λόγο στον κύριο Τάκουλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω τη μητρική μου, γιατί μερικά πράγματα μπορώ να τα πω καλύτερα στη μητρική μου γλώσσα. Λοιπόν, για αυτή την εκδήλωση ήμουνα στην ε, εκδήλωση αυτή ο αντιπρόεδρος ήθελε να εκφράσει ιδιαίτερα τις ευχαριστίες του γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετικοί και οι συνάδελφοι και η δουλειά που έκαναν και Θα ήθελα βεβαίως και εγώ να ε, εξ του να ευχαριστήσω ε, τους πάντες. Ε, βεβαίως θα, έρθω και εγώ στο σημείο αυτό. Αλλά πάμε στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των προηγούμενων ε, της 10ης Νοεμβρίου και της, 20, 20, και 23ης. Αν έχετε πρόβλημα να μου το πείτε μέχρι το τέλος της ε, Τη συνεδρίαση. Οι Ανακοινώσει του Προέδρου είναι μόνο η τα γλωσσικά. μπορείτε να μιλήσετε Ολλανδικά, δεν μπορείτε να ακούσετε Ολλανδικά, κατά τα λοιπά υπάρχουν διάφορες γλώσσες τι οποίε μπορείτε να μιλάτε αλλά όχι να ακούτε. Πάμε στην ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με την κυρία Ρέντινγκ. Πρόγραμμα για την Ιθαγένεια. Πραγματικά Όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία. Ξέρουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για το θέμα αυτό. Χαίρομαι που δεν έχουν άλλοι την ε, αρμοδιότητα για, το, για την ε, εκθέση αυτή, γιατί δεν κατάλαβα πώς χάθηκε το έτος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα της ηθαγένειας πάντα ήταν ε, δημοφιλές στην, στην Επιτροπή μας. Μιλούμε για τη δυνατότητα των πολιτών να μπορούν να συμμετέχουν στι δραστηριότητέ μα. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πολύ και με τον πολιτισμό και με την εκπαίδευση και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που έχουμε σήμερα αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Προς το παρόν, η κυρία Βερζιά κάνει μια νομοθετική πρόταση για το θέμα του Ευρωπαϊκού Έτους Ιθαγένειας 2013 και πραγματικά θα περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι θα μας πει η Επίτροπος Ρέντινγκ και τι έχει αναλάβει για το νέο αυτό πρόγραμμα. Παρακαλώ, Βιβία, να έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να παρουσιάσουμε την πρόταση της Κομισιόν για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους ε, πολίτες ε, 2014-2020. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα σας αναφέρω και κάποια πράγματα για τις ε, ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέονται βεβαίως με αυτό το θέμα. Καταρχάς θα σας πω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερο όνομα, καλύτερος τίτλος για αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Ευρώπη για τους πολίτες. λέει απλά αυτό ακριβώς που είναι η Ευρώπη. Και συνήθως το ξεχνούμε. Όταν μιλούμε για την Ευρώπη, μιλούμε για ελλείμματα, για τράπεζες, για α, μη βιώσιμες δαπάνες. Μιλούμε για το six-pack, το νομοθετικό. Μιλούμε για την ένωση των φορολογικών και οικονομικών πολιτικών. Αλλά δεν θυμόμαστε ότι ό,τι κάνουμε τελικά γίνεται για τους πολίτες. Για αυτά τα 500 εκατομμύρια πολιτών που βρίσκονται στον πυρήνα όλων των πολιτικών μας και ο λόγος ύπαρξης της Ευρώπης είναι ακριβώς αυτός. Να δώσει αυτή την χειραφέτηση στους πολίτες για να μπορούν να συμμετέχουν. Και αυτό ακριβώς κάνει και το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Αυτό λοιπόν ήταν που έπρεπε να επιλεγεί και αυτό επελέγει. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ε, Ευρώπης, τα προβλήματα που έχουμε που δεν είναι μόνο οικονομικά ή χρηματοδότησης, αλλά είναι και, θέματα, είναι και προβλήματα εμπιστοσύνης. Μπορούμε λοιπόν να τα αντιμετωπίσουμε μόνο αν έχουμε τους ε, πολίτες στο πλευρό μας. Αυτοί πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι δικά τους τα προγράμματα και ότι ανήκουν σε αυτά. Αν γνωρίζουν ότι εμείς, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν υπάρχουμε για να τους δίνουμε λύσεις και ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτές τις λύσεις, θα μπορούν και αυτοί να είναι περήφανοι που είναι Ευρωπαίοι, γιατί μας βοηθούν να δημιουργήσουμε αυτό το κοινό οικοδόμημα. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει αυτό το νέο εργαλείο, το, Ευρώπη, το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Καταρχάς να σας κάνω μια γενική παρουσίαση του προγράμματος και τι σημαίνει. Έχει δύο θεματικές ενότητες. Το ένα είναι η μνήμη και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια και το άλλο είναι η δημοκρατική δέσμευση και η συμμετοχή στα κοινά. Πρώτον, η πρώτη πτυχή έχει να κάνει με την ιστορία μας. Πρέπει να θυμόμαστε τα θύματα των απολυταρχικών καθεστώτων, του ναζισμού, του στελινισμού. Πρέπει να προωθήσουμε την ανοχή στις κοινωνίες μας. Αν δεν καταλάβουμε το παρελθόν μας, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε το μέλλον μας, δεν μπορούμε να, να ενοποιήσουμε την Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Και το, εσείς το κάνετε στις ε, εκλογικές σας περιφέρειες, εγώ το κάνω όπου μπορώ, όταν μιλώ με νέους. Και καταλαβαίνω ότι το να θυμόμαστε το παρελθόν δεν είναι δυστυχώς δεδομένο. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει αυτή η πτυχή της μνήμης. Η δεύτερη τώρα διάσταση, η δέσμευση και η συμμετοχή στα κοινά έχει να κάνει με την ενίσχυση της κατανόησης που έχουν οι πολίτες για το πώς λειτουργούν και πώς εκπονούνται οι ευρωπαϊκές πολιτικές στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Πώς ε, οι δράσεις τους συνδέονται με την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και πώς μπορούν να τους ε, βοηθήσουν να συμμετέχουν. Βεβαίως μιλώ κυρίως για τις ε, εκλογές, τις ευρωπαϊκές, τις ευρωεκλογές, στις οποίες, για τις οποίες θα πρέπει να συνεργαστούμε στους επόμενους μήνες για να υπάρξει ένα κοινό πρόγραμμα. Σε πλαίσια λοιπόν αυτής της, ναι, της δεύτερης διάστασης ε, μπορούν να χρηματοδοτηθούν διάφορα προγράμματα όπως ας πούμε συναντήσεις των πολιτών, προγράμματα της κοινωνίας των πολιτών, ε, προγράμματα αδεφοποίησης πόλεων. Μέσω λοιπόν όλων αυτών των γεγονότων τα, οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τις πολιτικές μας τον τρόπο με τον οποίο ε, εκφωνούνται και λαμβάνονται οι αποφάσεις και που δεν είναι απλός, πώς λειτουργεί το σύστημα και ποιες είναι οι συνέπειες όλων αυτών των προγραμμάτων και της, ε, όλης αυτής της διαδικασίας στην καθημερινή του ζωή. Όλα αυτά τα προγράμματα βεβαίως πρέπει να έχουν και μια πτυχή υπερεθνική, μια διάσταση ευρωπαϊκή και βεβαίως θα υπάρχει και μια τρίτη οριζόντια διάσταση, η οποία θα αφορά και τα δύο, και τις δύο θεματικές ενότητες, και αυτή που αφορά την ιστορική μας μνήμη και αυτή που αφορά την συμμετοχική. Τα προγράμματα θα ε, εξετάζονται μέσω ε, αξιολογήσεων ομοτήμων, μέσω καινοτόμων ε, προγραμμάτων και ιδεών θα κοινοποιούνται παντού και αυτό θα μπορέσει να δημιουργήσει καλύτερες υποδομές, καλύτερες δυνατότητες ώστε να μάθουμε από τις εμπειρίες μας και να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις επενδύσεις μας. Τώρα, ποιος μπορεί να, να κάνει αίτηση για αυτή την χρηματοδότηση. Το προγράμματα αυτά είναι ανοιχτά για οργανώσεις που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και που έχουν ε, υπερεθνική διάσταση, ας πούμε τοπικές αρχές, ερευνητικέ ομάδες, think tanks, ομάδες πολιτών, ή άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και υπάρχει μια απόλυτη συνέχεια στα υπάρχοντα προγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανώσεις που ήδη συμμετέχουν σήμερα μπορούν να ξανασυμμετέχουν και στο μέλλον. Τρίτον είναι η διαχείριση και ο προϋπολογισμός. Θα υπάρξουν ε, βεβαίω κάποια δάνεια ε, δράσης και δάνεια επιχειρησιακά, θα υπάρξουν κάποιες συμβάσεις. Ε, θα υπάρξει μια εκτελεστική υπηρεσία η οποία θα διανύμει όλα αυτά τα κονδύλια που σημαίνει ότι θα υπάρξουν εξοικονομήσεις και τώρα μιλώντας για χρήματα το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες έχει μια πρικοδότηση 229 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορώ να πω ότι μιλούμε για αύξηση 15 εκατομμυρίων. Δεν είναι πολλά, αλλά δεν είναι και αμεληταία. Γιατί τα έχουμε αναδιοργανώσει, που σημαίνει ότι αυτά τα λίγα χρήματα θα έχουν πολλές ε, συνέπειες, γιατί το πρόγραμμα είναι πιο στοχοθετημένο προς τα αποτελέσματα και πιο φιλικό προς το χρήστη. Επομένω είναι και πιο αποδοτικό προς τα ε, οικονομικά του. Ε, και είμαι σίγουρη ότι θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα αποτελέσματα που θα είχε ο ίδιος, το ίδιο αυτό ποσό για προγράμματα που τρέχουν τώρα. Εφόσον θέλουμε λοιπόν να έχουμε τέτοια, ποσά πρέπει να έχουμε και καλές ιδέες. Η δική μου πρόθεση ώστε αυτά τα ε, χρήματα να έχουν όντως αποτέλεσμα, είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν ε, εταιρικέ σχέσεις. Πρέπει να έχουμε ε, σωστούς καλού εταίρου όταν προσπαθούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να γνωστοποιήσουμε και στους πολίτες τι ακριβώς γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι το σύστημα δεν ξεκινάει από πάνω προ τα κάτω, αλλά από κάτω προ τα πάνω. Και εκεί βεβαίω χρειάζεται και η βοήθεια των Ευρωβουλευτών να αναλάβουν και αυτή την ευθύνη που του αναλογεί, να πάνε στου πολίτε και να χρησιμοποιήσουν ε, τα μέσα που του δίνεται και να δεσμεύσουν, να, να προσελκύσουν του πολίτε. Υπάρχει ήδη μια έκθεση για την επικοινωνία, την οποία σας είπα ότι θα σα αναφέρω. Πριν το κάνω, θα ήθελα να σας πω τα σημερινά νέα. Στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας έχουμε νέο Γενικό Διευθυντή. Μπορεί να μην εκπλαγείτε όταν ακούσετε το όνομα, γιατί είναι παλιός φίλος. Ο Γκρέγορη Πόλτσε. Εκεί είναι, τον βλέπετε. Διορίστηκε από το κολέγιο σήμερα το πρωί. Η πρώτη του δραστηριότητα τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά είναι να έρθει σε αυτή την Επιτροπή. Χαίρομαι που σας έχουμε σήμερα εδώ, Γκρέγκορη. Από εδώ και μπρος, λοιπόν, ο Γκρέγκορη θα είναι ο άμεσος συνομιλητής σας για όλα όσα αφορούν την επικοινωνία. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε στον τομέα της επικοινωνίας. πρέπει να κάνουμε κάθε άλλο παρά να, πρέπει να κάνουμε τα πάντα ε, πλην του να μιλούμε μόνο για την επικοινωνία. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών εξ ονόματος των οποίων μιλούμε. Τι κάνει η Ευρώπη, πώς συμβάλλει για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Αυτή είναι η προσέγγιση της επικοινωνίας. Υπάρχουν τρία πολλά, πολύ απλά σημεία. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε την ε, ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τις ε, ευκαιρίες που τους προσφέρει η Ευρώπη. Δεύτερον, η επικοινωνία είναι εργαλείο που φέρνει, που διαβιβάζει μηνύματα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους δημοσιογράφους, πρέπει να βοηθήσουμε τους μιμι, τα ΜΜΕ για να μπορέσουν να έχουν το υλικό που τους χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να μεταδώσουν το μήνυμα. Και τρίτον, πρέπει οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση. Να σας πω λοιπόν κάποια πράγματα για τις τρεις αυτές πτυχές. Καταρχάς, αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις ευκαιρίε που δίνει η ενιαία αγορά. Παρόλο που δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, γιατί μόνο, μονίμως μιλούμε για την ενιαία αγορά. Μιλούμε, θα έπρεπε να μιλούμε για τον κοινό μας χώρο, γιατί η Ευρώπη είναι το, πολλά περισσότερα από μια αγορά. Είναι ένα μέρος που ζούμε, είναι το μέρος που υπάρχουμε, είναι το μέρος που ανταλλάσσουμε ιδέες, που επικοινωνούμε. Έχω υιοθετήσει λοιπόν την πρώτη έκθεση για την Ιθαγένεια, κάτι που έγινε τον Οκτώβριο του 2010. Και εκεί απαντώ στο αίτημα που είχε, κάνει το, που είχε υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να δούμε δηλαδή α, ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ποια είναι τα σχόλια που έχουν να κάνουν, ποια είναι η κριτική που έχουν να ασκήσουν και επίσης τι ε, τους ενδιαφέρει, τι είναι σημαντικό ως ιδιώτες, ως καταναλωτές, ως φοιτητές, ως επικελματίες ή ως ενεργοί πολίτες. Η έκθεση λοιπόν έδειξε ότι υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης και αυτό ήταν ένα από τα βασικά εμπόδια. Ε, πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν ποιε είναι οι ευκαιρίε που του δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ποια είναι τα ωφέλη αυτή τη ε, ε, υπήρου, ούτε ποια είναι τα ωφέλη του να έχει κανείς την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και γι' αυτό, σε αυτή την έκθεση, έχω καταγράψει πέντε δράσεις τις οποίες ε, θα, με τις οποίες θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση κομισιών. Μία από αυτές, και το είπατε πρόεδρε, είναι η πρότασή μου του Αυγούστου 2011, ώστε το 2013 να γίνει το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Μόλις εγκριθεί αυτό από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα γίνει μια στοχοθετημένη ε, ενημερωτική εκστρατεία με πολλές αποκεντρωμένες δράσεις οι οποίες θα γίνονται και σε εθνικό και σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις με τους πολίτες, να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε γιατί πολλά από τα ερωτήματα για τα οποία υπάρχουν ήδη α, ε, απαντήσεις δεν τα γνωρίζουν. Ε, αυτό το ευρωπαϊκό έτος λοιπόν νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση να βάλουμε τους ε, πολίτες στην ε, καρδιά, στον πυρήνα της πολιτικής ατζέντα και εσείς θα μπορέσετε να βοηθήσετε. Βεβαίω αυτό το έτος θα είναι ε, ένα έτος πριν από τις ευρωεκλογέ. Θα είναι λοιπόν κρίσιμο έτος γιατί ακόμα δεν θα είμαστε σε εκστρατεία εκλογική και ακόμα θα μπορούμε να, εξηγούμε με αντικειμενικό τρόπο τι κάνει η Ευρώπη για τους πολίτες της και θα μπορούμε να βασιστούμε σε όλα αυτά για να κινητοποιήσουμε το εκλογικό σώμα για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τις ζωές των πολιτών και να τους δείξουμε ποιες είναι οι δράσεις και που εμείς και οι, τις, ε, Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ποιες είναι οι δράσεις που έχουν αναλάβει. Βεβαίως περιμένω ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα συμμεριστούν την πρωτοβουλία αυτή και θα πάρουν μέρος στο διάλογο. Δεύτερο, η επικοινωνία ως αποτελεσματικό εργαλείο για να μεταδοθούν τα μηνύματα από και προς τα ΜΜΕ. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές είναι κάτι που ως μέλος Εθνικού Κοινοβουλίου αλλά και ως δημοσιογράφος για πάνω από 20 χρόνια, το έχω ζήσει πολύ και το πιστεύω. Η επικοινωνία δεν είναι ο σκοπός, είναι το εργαλείο. Ένα εργαλείο που, βοηθάει να ε, γίνουν πραγματικότητα οι πολιτικές. Αν δεν υπάρχει καλό μήνυμα, η επικοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει λοιπόν πρώτα να βρούμε ποιο είναι το μήνυμα και μετά να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα ώστε να περάσει αυτό το μήνυμα. Μπορούμε λοιπόν να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε για κάτι, για κάτι συγκεκριμένο, για δράσεις, για ουσία, για πολιτικές και αυτό είναι αυτό που θα μας βοηθήσουν να, που να κάνουμε τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Προφανώς δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με όλους και τον καθένα ξεχωριστά, τους πολίτες μας. Γι' αυτό χρειάζεται να, κάποιος να μας βοηθήσει για να πολλαπλασιαστεί το μήνυμα. Και χρειαζόμαστε τα ΜΜΕ και τα ΜΜΕ χρειάζονται εμάς για να τους δώσουμε το υλικό. Και μετά, ό,τι τους δώσουμε, με βάση την ε, ελευθερία του τύπου και της έκφρασης, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Γι' αυτό λοιπόν ε, υποστηρίζουμε την εκπαίδευση των, ε, ε, των δημοσιογράφων, όπως αναφέρεται και στην έκθεση Locking για, τον, για τη δημοσιογραφία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Πρέπει να δώσουμε κάποια εργαλεία, κάποια μέσα, σε, ακόμη και σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν ήδη. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να ξέρουν από πού να πάρουν πληροφορίες, από πού να ενημερωθούν. Επίσης, όπως λέει η έκθεσή σας, ενίσχυσα την στήριξη που δίδεται στο Euronews για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι ένα μοντέλο ανεξάρτητης αντικειμενικής ποιοτικής ε, δημοσιογραφίας, τηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Με την ε, στήριξη αυτή το Euronews έχει ανοίξει ένα γραφείο εδώ στα, στις Βρυξέλλες για να είναι πιο κοντά στην καθημερινή ε, δουλειά των ε, Ευρωβουλευτών ε, και, των, ε, και στην Κομισιόν για να καλύπτει γενικώ τα ευρωπαϊκά γεγονότα. Και θα ήθελα να σας ε, καλέσω όλους να πάτε στο γραφείο του Euronews και να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα με, πιο, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να έρθετε και εσείς σε επαφή μέσω του Euronews με τους πολίτες σας. Και επίσης, κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, το Euronews ήταν ε, διαθέσιμο και στα πολωνικά για πρώτη φορά ως πιλωτικό πρόγραμμα. Βεβαίω πρέπει να αναλύσουμε το, την διαδικασία αυτή, δεν μπορούμε να σα δώσουμε ακόμα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι καταρχά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και μιλώντα για τι γλώσσες, ξέρετε ότι το Euronews είναι πολύγλωσσο, ε, εκπέμπει και στα αραβικά και στα φαρσί. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω σε εσά γιατί είναι σημαντικό αυτό. Οι εταίροι στην ε, ε, Μεσόγειο είναι εξίσου σημαντική και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το Euronews με αυτόν τον τρόπο. Η ενίσχυση λοιπόν του Euronews ήταν ένα, μία από τις δράσεις που προέκυψαν από την έκθεση και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την πολυγλωσία αυτή και οι ευρωβουλευτές θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα. Κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα εφόσον το επιθυμείτε κι εσείς. Και επίσης, η άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση, σε ενημέρωση για τους πολίτες. Κυρίως όταν έχουμε φοιτητές αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. μα. λένε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, αλλά εγώ αυτέ τις πληροφορίες που μπορώ να τις βρω. Βασίστηκα λοιπόν ε, στην ε, εταιρική σχέση που έχουμε με το, ε, με το κέντρο επικοινωνίας του Europe Direct και το δίκτυο Europe Direct και έχουμε τώρα 487 κέντρα ενημέρωσης του Europe Direct που επικοινωνούν άμεσα με τους πολίτες μας. Μιλούν οι εργαζόμενοι εκεί την γλώσσα της χώρας, έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και μπορούν να περάσουν το μήνυμα και να επικοινωνήσουν με τους πολίτες. Είναι πολύ αποτελεσματικό το Europe Direct και βεβαίως μιλώντας για τη νέα γενιά έχουμε και, το, και τα μέσα του ίντερνετ. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστοσελίδες και τα λοιπά που μπορεί κανείς να μπει και να πάρει πληροφορίες. Ζήτησα λοιπόν από την υπηρεσία μου να δημιουργήσει μία, ε, μία πύλη, μία θηρίδα ενιαία όπου θα μπορεί κανείς να μπαίνει και μετά να, και θα βρίσκει τις πληροφορίες που θέλει μέσα από την κεντρική πύλη. Πάντα μιλούμε για την νεολαία. Η νεολαία όμως δεν είναι μία συμπαγής ομάδα. Υπάρχουν τεράστιες ε, διαφορές μεταξύ ε, φοιτητών και 15χρονων παιδιών. Ε, αν λοιπόν δεν ξεκινήσουμε από τα παιδιά, πώς θα φτάσουμε στους εφήβους. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και μια ειδική ιστοσελίδα, την γωνιά των παιδιών, που είναι αφιερωμένη σε μικρά παιδιά και που θα βγει online αύριο. Και πρόεδρε, αν θέλετε, ευχαρίστως να σας κάνω και μία παρουσίαση αρχές του επόμενου έτους για το Kids Corner, για τη γωνιά των παιδιών. Ωραία. Η ιστοσελίδα λοιπόν αυτή δεν είναι προφανώς τέλεια. Θέλω και εγώ τη δική σας συμβολή για να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Αλλά έχει να κάνει με την ενημέρωση για τα δικαιώματα των παιδιών. Γιατί τα δικαιώματα των παιδιών είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της Κομισιόν. Έχει να κάνει με παιχνίδια, με κουίζ, με πληροφορίες για την Ευρώπη. Με, και είναι γραμμένα όλα αυτά με έναν τρόπο που τα παιδιά ελπίζουμε ότι μπορούν να τον καταλάβουν για να μπορούν να μάθουν, να παίζοντας για την ε, σημασία της Ευρώπης. Οπότε, αν μπορείτε, μπείτε να δείτε την ιστοσελίδα και αν μπορείτε να μου δώσετε και την συμβολή σας, θα σας ήμουν ευγνώμων. Ίσως να μπορούσατε να το δείτε και με εμπειρογνώμονες που έχετε στους, ε, στις εκλογικές σας περιφέρειες, για να σας πούνε και αυτοί τι είναι καλό και τι όχι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ιστοσελίδα, να την τροποποιήσουμε. Καταλαβαίνετε νομίζω ότι προτίθεμαι να κάνω. Θέλω να γίνουν τα πράγματα συγκεκριμένα. Θέλω να είμαστε πρακτικοί. Και αυτά είναι καινούργια στοιχεία βέβαια. Όλα τα παλιά προγράμματα εξακολουθούν να τρέχουν. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Να πω απλώς Κυρία Πρόεδρε, δύο πράγματα για τα λεφτά, για τα χρήματα. Άκουσα το, αυτό που λέτε. Έχετε περίπου 8 εκατομμύρια σε απόθεμα για την κοινοποίηση της Κομισιόν για τον Προπολογισμό 2012. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κάποιες επιλογές. Οι υπηρεσίε τη ε, Γενική Διεύθυνση ε, Επικοινωνία έχουν ε, αποστείλει σε εσά πολλά έγγραφα και εξηγήσει. Και τώρα έχετε και τον Γκρέγκορη. Και θα είναι στη διάθεσή σα για να σας απαντήσει σε ό,τι ερωτήματα έχετε. Ένα από τα αιτήματά σας ήταν ότι θέλετε να ε, το Euronet, το πρόγραμμα. Επιμείνατε πολύ σε αυτό. Κάναμε μια ανάλυση. Δεν ήταν πολύ ικανοποιητικά τα πράγματα, αλλά προσπαθούμε να πιέσουμε ώστε να βελτιωθεί το πρόγραμμα, να είναι πιο αποτελεσματικό. Θα επιμηκυνθεί λοιπόν. Βεβαίως έχουμε και τα 8 εκατομμύρια που λείπουν, οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που θα πρέπει ίσως να διακοπούν. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε από κοινού γιατί είναι κοινή μας ευθύνη. Νομίζω αρκετά μίλησα κυρία Πρόεδρε, οπότε ευχαρίστω να ακούσω ερωτήματα και να σας απαντήσω. So, thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν συνεχίσουμε, έχουμε πρόβλημα με τα γερμανικά στη Διερμηνία. Οι Γερμανοί θα μιλήσουν ελληνικά ή θα πρέπει να σταματήσουμε για λίγο για να ε, συνεχίσει διορθωθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Κάβαντα, ο οποίος θα μιλήσει γαλλικά φαντάζομαι. Θα προσπαθήσω να μιλήσω γαλλικά. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Επίτροπο, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύο πολύ ξεκάθαρα πράγματα σε σχέση με την ε, πρωτοβουλία αυτή για το έτος της ε, υπηκότητας, το έτος της ηθαγένειας. Αυτό το οποίο είπατε για τα μέσα ενημέρωσης που θα εκπλήξουν μόνοι όσους δεν γνωρίζουν την υπόθεση είναι πολύ ευπρόσδεκτα. Και τέλος χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνει προτεραιότητα στο μοναδικό κανάλι που διαθέτει η Κομισιόν εδώ και πολλά χρόνια, το Euronews. Χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι μια επιχείρηση που τη γνωρίζω επαγγελματικά, είναι καλού επίπεδου, έχει περιορισμένε δαπάνες, εργάζεται καλά, είναι πολύγλωση και ασχολείται με τα θέματα, τα κοινοτικά, ευρωπαϊκά κοινοτικά, ξεπερνά τα εθνικά και μάλιστα σε πολλές γλώσσες, πράγμα που είναι απαραίτητο. Πιστεύω ότι θα πρέπει το επαρθμό, το Euronews να γίνει το ανεξάρτητο όργανο. Φυσικά επιδοτείται. Εμείς οφείλουμε, κυρία Επίτροπε, και εμείς οι ίδιοι να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του καναλιού αρκεί να παρατηρήσει κανείς ότι καλύπτει σχεδόν το σύνολο της ε, κοινότητας. Ε, σας ευχαριστούμε λοιπόν που θέσατε το δάχτυλο επί ενός θέματος σωστού και υψηλής ποιότητας. Το πρώτο μέρος της ε, παρουσίασής σας αναφερθήκατε στο καθήκον για την μνήμη και την ιστορία δεν νομίζω ότι μπορούμε να επικρίνουμε αυτή την πρότασή σας, είναι επιβαλόμενη, αλλά ε, σε μια στιγμή που η Ευρώπη συζητά τα θεμελιώδη θέματά της και που έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη εποχή, τον χρηματοοικονομικό πόλεμο στον οποίο ζούμε παγκοσμίω, η πρωτοβουλία αυτή είναι αξιόλογη και πρέπει να γίνει πιο εμφανής. Το λέω αυτό γιατί θα ήθελα επιτέλους οι Δυτικοευρωπαίοι, οι οποίοι δεν έχουν αρκετούς ήρωες, τους ιδρυτές, τους απελευθερωτές της Γερμανίας κλπ. Θα ήθελα να θυμηθεί ότι στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έγιναν παρόμοια πράγματα και ότι αυτά δεν είναι παρκώς γνωστά. Θα ήθελα να ε, θυμίσω τους ήρωες του 48 στην Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία και ακόμα λίγο νωρίτερα τις ε, εξαιρετικά θαραλέες πράξεις ενός 22χρονου πρόεδρο των φοιτητών της Βουδαπέστης, του Ζωέλ Μπραντς, ο οποίος έσωσε Εβραίους από τα φορτηγά, εκατοντάδες χιλιάδες. Θα πρέπει να είναι γνωστό το όνομα της κυρίας Γκουζι Φλάισμαν, μιας ηρωίδας από την Πρατισλάβα, η οποία ε, ξόδεψε την περιουσία του ε, συζύγου της που ήταν βιομήχανος, όπως την λίστα του Σίγκλερ, για να σώσει ανθρώπους. Ανέβηκε στο φορτηγό με τα τελευταία μικρά παιδιά της γειτονιάς της και πήγε και χάθηκε. Θα ήθελα να θυμόμαστε το παρελθόν που θα μας δώσει το μέλλον. Παρότι αυτό προέρχεται από έναν, μια περίοδο Μαρέ και Ντόλμαν, μία από τους τρεις επιζήσαντες ε, ε, του γκέτου της Βαρσοβίας, ε, μεγάλη, μια μεγάλη καρδιολόγος από τη Βαρσοβία με τον Κεμέκ και τον Βαλέσα. Έτμοντ Μπάουνκα, ηλεκτρολόγος στο Γκτάνσκ, που ήταν ο προκάτοχος του Βαλέσα θα έλεγα. Στο, στο πάνθεον αυτό θα πρέπει να υπάρχει ο γιαν παλαν Παλάν, ένας 22χρονος φοιτητής, ο οποίος ε, στη, το 1968 αυτοπυρπολήθηκε θα υπάρχουν ο, καρδινά, ο και το καρδινάλης Βυσίνσκι από το 68 στην Πολωνία. Αυτοί που έδωσαν τη δύναμη στους καθολικούς της Πολωνίας να ρίξουν το κομμουνιστικό καθεστώς. Θα ήθελα να θυμόμαστε τον Ντούπτσεκ, να γνωρίσουμε για την άγνωστος τον Ήρη Πέλικαν, τον θαραλέο Γενικό Διευθυντή της ε, ραδιοτηλεόρασης της Τσεχοσλοβακίας, ο οποίος ε, διέφυγε από τη χώρα του κυνηγημένος από την αστυνομία γιατί επί τρεις μήνες ε, μετέδιδε ανεξάρτητες εκπομπές και άλλους. Είναι στιγμή πλέον, ήρθε η κατάλληλη στιγμή, κυρία Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, να φτιάξουμε, να παρουσιάσουμε αυτούς τους γνωστούς και αγνώστους ήρωες της Ευρώπης που έφτιαξαν την εποχή στην οποία ζούμε. Ευχαριστώ. Θέλω να πω στους συναδέλφους ότι η κυρία Επίτροπος θα μείνει εδώ μέχρι τις 4.30. Ε, ξέχασα να σας το πει από την αρχή. Ζητώ συγγνώμη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε, αλλά πρέπει να ε, κάνουμε οικονομία στο χρόνο. Κύριε Κουρία. Ε, λειτουργεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα μετά από όσα άκουσα από την κυρία Ρέντινγκ, ιδιαίτερα λόγω της ε, αντίληψης ε, το να μιλάμε για μια Ευρώπη που δεν αποτελείται μόνο από μια αγορά ότι θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τους πολίτες και όχι για, μόνο για λόγους οικονομικούς ή χρηματοπιστωτικούς και την κρίση που αντιμετωπίζουμε και αυτά είναι πράγματα τα οποία μας ε, δείχνουν πώς θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν στους Ευρωπαίους και τους πολίτες. Χαίρομαι λοιπόν που άκουσα αυτή τα, αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα μέσα από την πρόταση της ε, Επιτρόπου. <clears throat> Πριν από μερικές μέρες, ό,τι φορά τη μνήμη, κάναμε μια ακρόαση αναφορικά με το θέμα των ολοκληρωτισμών στην Ευρώπη για τα εγκλήματά τους ε, και πολλοί συνάδελφοι πολλές οργανώσεις μας ε, μίλησαν για το πώς ε, θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το γεγονός και που δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας, αλλά και την προσοχή που αποδίδεται στον εξυγχρονισμό με όλων των μέτρων που υπάρχουν και το μέσο που υπάρχουν στην επικοινωνία. Ήθελα απλά να υπογραμμίσω το εξής, ε, δρατώμενο της ευκαιρίας που παρίσταται ο νέο Γενικό Διευθυντή, τον οποίο και συγχαίρω για τον ε, διορισμό του, την απλούστευση, την απλοποίηση, για να μπορέσουν να συμμετέχουν οι πολίτες και οι οργανώσεις ε, στο πρόγραμμα αυτό. Διότι ειδικά σε ό,τι φορά αυτό το πρόγραμμα μιλάμε για ενώσεις, για πολίτες, για οργανώσεις μικρές, μικρών, μικρού μεγέθους που δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικούς φραγμούς για να έχουν πρόσβαση στα στους πόρους του προγράμματος. Για ό,τι άκουσα αυτοί αυξήθηκαν αν και όχι ουσιαστικά, αλλά είναι ένα σημαντικό μήνυμα σε περίοδους κρίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι η Κομισιόν και τα γραφεία της, νέου προγραμματισμού θα μπορούσαν να σκεφτούν να έχουν λιγότερα έγγραφα και να αποδώσουν μεγαλύτερη προσοχή στο περιεχόμενο που ενδιαφέρει και ιδιαίτερα τους πολίτες. Ευχαριστώ. Μετά από αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε δύο λεπτά διάλειμμα για να ξαναξεκινήσει το σύστημα. Οπότε προς το παρόν θα πρέπει να κάνουν υπομονή οι Γερμανοί. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστώ την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Να πω επίσης ότι για να προσεγγίσουμε τους πολίτες ε, θα πρέπει να ε, καταστήσουμε γνωστό τι κάνει η Ευρώπη για τους πολίτες και ποια είναι η Ευρώπη την οποία ε, απεργαζόμεθα. Ε, θεωρώ ότι μάλλον σήμερα το πρωί είχα συνάντηση με μια ομάδα πολιτών και όταν τους είπα το 70% περίπου όλων των, όλης των Ισπανικών αλλά και των αυτονομιών στην ε, Ισπανία προέρχονται από την Ευρώπη εξεπλάγησαν, δεν πιστεύουν στα αρθιά τους διότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θεωρώ ότι αυτή η συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι πολύ σημαντική. Τώρα βρισκόμαστε γύρω στους, είμαστε περίπου 790 βουλευτές με τους καινούριους που έφτασαν. Δεν είμαστε τόσοι πολλοί, και, θεωρούμε ότι 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που, στους οποίους εκπροσωπούμε, συμπεριλαμβανομένου και του κύρου, του γοήτρου που έχει η Ευρώπη, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, στην ουσία το κόστος αναπολίτη των ευρωπαϊκών θεσμών είναι 3 ευρώ αετησίως θεωρώ ότι αυτές οι λεπτομέρειες θα πρέπει να τις γνωστοποιήσουμε. Θα πρέπει να δείξουμε ποια είναι η πραγματικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κομισιόν και τις επιπτώσεις του στην ζωή των πολιτών. Ε, έχουμε οργανώσει το παρλαμεντάριο κάτι το οποίο εξηγεί πολύ σωστά την ε, ιστορία της Ευρώπης. Όταν μιλάμε για τον τύπο, θα πω ότι πρέπει να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια στον εξειδικευμένο τύπο, στον οικονομικό τύπο, τον αθλητικό τύπο, τον ε, πολιτιστικό τύπο. Δηλαδή τα εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης είναι ενδιαφέρον να, μάλλον πρέπει να τους ζητήσουμε να ασχοληθούν λίγο παραπάνω με τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Συγχαρητήρια στον κύριο Πόρτσα, τον ε, νέο Γενικό Διευθυντή. Συγχαρητήρια λοιπόν ε, κύριε Γενικέ. Τρία πράγματα θα ήθελα να θίξω. Πρώτον, άκουσα για το εντύπαρ και το Euronews, το Euronews είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και πέρα από το Euronews, το μιλάμε για επικοινωνία, διότι οι πολίτες ε, πρέπει να ακούνε και το τι συμβαίνει σε επίπεδο κρατών ε, μελών ε, στην Ένωση και μέσω των εθνικών μέσων ενημέρωσης ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το ζήτημα διότι ε, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν το τι συμβαίνει στην ε, Ευρώπη και όχι μόνο στις Βρυξέλλες. Οι πολλοί πολίτες ε, δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα, δεν έχουν ιδέα Ακόμα και οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι του BBC έχουν άγνοια πολλών θεμάτων. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και στα άλλα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν να διασφαλίσουμε πως οι πολίτες θα έχουν, έχουν καλύτερη ιδέα για το πώς λειτουργούμε, τι ακριβώς κάνουμε, σε τι χρησιμεύουμε. Ε, και αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και άμεσα θα έλεγα να ε, υπάρχει ενημέρωση και στα σχολιά. Εμείς ε, ως ε, αρμόδια επιτροπή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες δυνατότητες τουλάχιστον να μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει, πώς λειτουργεί, τι προσφέρει. Θα ήταν χρήσιμο εάν το πετυχαίναμε. Όσα είπατε για το διαδίκτυο, για την πύλη κλπ. είναι πολύ ωραία. Πρέπει να τα προωθήσουμε, πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Αλλά χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι την επικοινωνία την ε, βλέπουν ε, οι πολίτες διαφορετικά από κράτος σε κράτος. Και θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν τους προκειμένου να ενημερωθούν. Ο κύριο Τάκουλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, μερικές σκέψεις επί του προγράμματος Ευρώπη των πολιτών που μου είναι αρκετά οικείο ως ε, εισηγητής, ε, θα θέλω να πω ότι πρόκειται για μια success story. Για ποικίλους λόγους, ο κ. Καβαντά αναφέρθηκε στους μεγάλους ε, Ευρωπαίους, αλλά εάν λάβουμε υπόψη την ευρωπαϊκή κληρονομιά, μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και την Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί πολίτες αυτών των περιοχών που αναφέρθηκαν προλίγου και για μένα αυτό αποτελεί μια επιτυχή ιστορία, επιτυχημένη ιστορία, success story. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτήν την ιστορική μνήμη της Ευρώπης και ενδεχόμενα να την ενισχύσουμε. Θα προτιμούσα να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια διαθέσιμα, ακόμα και αν το ποσό αυξήθηκε κατά τι, διότι Υπάρχουν κάποια σχέδια σημαντικότατα, ε, σχέδια bottom-up, όπως είπατε, και αυτό είναι ο λόγος ε, για τον οποίο σήμερα έχουμε αυτά τα διαθέσιμα κονδύλια. Ε, να πω επίσης ότι δεν έχω να παραδείσω πολλά στα λεγόμενα της Επιτρόπου. Θα θέλαμε να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και αυτό σε όλα τα επίπεδα, αλλά και μία παρατήρηση να κάνω. Αυτές οι ομάδες ε, προβληματισμού που καλύπτονται από το πρόγραμμα, ορισμένοι μιλούν για ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά ίσως ε, θα έπρεπε να δώσουμε και μία ευκαιρία στους ε, νέους ε, πρωταγωνιστές, ε, να έχουμε νέα άτομα, νέα όργανα τα οποία θα συνεργαστούν μαζί μας και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και Πρόεδρε, διερωτώ με πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε περαιτέρω τους πολίτες. Ξέρουμε ότι η περίοδος είναι δύσκολη με την ε, οικονομική κρίση που διανύουμε και ακούγεται ότι η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη προς τις αγορές και πως ε, οι αγορές ε, έχουν μπει στο επίκεντρο της Ευρώπης και δεν υπάρχει μια κουλτούρα της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και του ευρωπαίου πολίτη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να περάσει αυτό το μήνυμα στους ε, πολίτες, να μιλήσουμε για τις ευρωπαϊκές ρίζες μας, για αυτό τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ευρωπαϊκή κληρονομιά και να καταστήσουμε ορατό ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από την κοινή αγορά ή τις οικονομικές ε, πολιτικές. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Επίτροπος τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η μνήμη. Η στοχοθέτηση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μπορεί να ενισχυθεί μέσω της μνήμης. Ο κύριος Καβαντά ανέφερε κάποια παραδείγματα από το παρελθόν. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω κι εγώ τα... την αναφορά αυτή. Πριν από 24 χρόνια α, απελευθερώθηκε τη Μισοάρα στην Ρουμανία και αποτέλεσε την πρώτη ελεύθερη πόλη της Ρουμανίας. Θυμάμαι ακόμα τους εορτασμούς όταν έπεσε ο Τσαουσέσκου, όταν άνοιξαν τα σύνορα, όταν ήρθαν οι Ευρωπαίοι, άνθρωποι από την ε, Ουγγαρία ήρθαν και έδειξαν την ε, αλληλεγγύη τους. Είδαμε λοιπόν την ε, αλληλεγγύη των πολιτών τότε. Τι θέλω να πω. Μεταξύ Ανατολής και Δύσης υπήρχε ε, το ε, τείχος του Βερολίνου πιο πριν το σιδηρούν παραπέτασμα. Νομίζω ότι οι χώρες των ανατολικών χωρών της Ευρώπης, των πρώην κομμουνιστικών χωρών, ε, δεν έχουν την αίσθηση ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Ας πάρουμε ας πούμε έναν, ε, ε, έναν Ρωμά. Δεν έχει την, την πεποίθηση ότι είναι Ευρωπαίος πολίτης. Μια φιλανδική αντιπροσωπεία πήγε στην πόλη μου στην Ρουμανία και επισκέφθηκε πληθυσμούς Ρωμά. Εμείς πήγαμε την τον προηγούμενη μέρα και δώσαμε δώρα στα παιδιά. Ε, το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει τη στρατηγική για τους Ρωμά. Σας ανέφερα πόσο καλό είναι ότι υπάρχει αυτή η στρατηγική και αυτή η στρατηγική πρέπει να, να εφαρμοστεί προς όφελος των πολιτών. Αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, ότι μεταξύ Ανατολής και Δύσης Πρέπει να υπάρξει προσέγγιση, πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη σε ανθρώπινο επίπεδο. Υπήρχαν και τα σύνορα Ουκρανίας-Σλοβακίας ε, και δεν μπορούσε κανένας να περάσει. Έπρεπε κανένας να, ταξιδέψει 150 χιλιόμετρα για να μπορέσει να πάρει μια άδεια για να περάσει. Τον καιρό του Τσεουσέσκου καταργήθηκαν οι κεραίες τηλεόρασης. Για να μην μπορούμε να ακούμε τις ομιλίες του Χάβελ. Ε, όλα αυτά πρέπει να, τα, ε, πρέπει να τα γεφυρώσουμε. Αυτό σημαίνει ενοποίηση και γι' αυτό πραγματικά χαιρετίζω αυτό το πρόγραμμα. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα συμμετέχουμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει κάποια πράγματα. Άκουσα τα διάφορα μηνύματα των συναδέλφων ε, και να πω ότι συχνά υπάρχει ε, αντίφαση μεταξύ του να λέμε και να κάνουμε. Είμαι εισηγήτρια για το ζήτημα της εισαγένειας ε, και να πω ότι όλοι συμφωνούμε στην αίθουσα αυτή τουλάχιστον ότι η ηθαγένεια δεν περιορίζεται μόνο στο δικαίωμα του εκλέγην, αλλά ούτε και στην αναγνώριση των δικαιωμάτων, όπως είπατε πολύ σωστά. Δεν πρόκειται για top-down, πρόκειται για bottom-up. Καντάντι ανάντι. Λοιπόν, ε, δεν θα να βασιζόμαστε μόνο στα άρθρα 20 και 21 τις συνθήκες, διότι αυτό κατ' εμέ αποτελεί άρνηση της ε, πολιτιστικής ταυτότητας της Θαγένειας ε, που για μας ε, και θέλω να προδικάσω τη συζήτηση διότι νομίζω ότι σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχαμε τους σκιώδης ηγητές για μας είναι πολύ ουσιώδης διάσταση. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ένα-δυο στοιχεία τα οποία ανάπτυξαν κάποιοι συνάδελφοι, η πολιτιστική και εκπαιδευτική διάσταση πράγματι είναι να δώσουμε τα μέσα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, να σταθούν πολίτες από την πιο τρυφερή ηλικία, δηλαδή να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου οι νέοι Ευρωπαίοι να μάθουν την ιστορία των κρατών της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, το νωρίτερο δυνατόν. Και αυτό δεν θα πρέπει να είναι ε, διάφορα προγράμματα αποκομμένα το ένα από το άλλο. Τώρα για τις επένδυτες πρακτικές και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε περαιτέρω, να αξιολογήσουμε ότι είναι καλό στον τομέα, ιδιαίτερα στα πολιτιστικά δίκτυα. Μα είπατε επίση ότι δεν υπάρχει επικοινωνία δίχω μήνυμα. Το μήνυμα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπλοκο σε αυτή την περίοδο τη ε, οικονομική κρίση και ο ρόλο των κρατών μελών ε, θα πρέπει να τονιστεί περαιτέρω. Στην ε, ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας και συγγνώμη που το επιμένω, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη, μισό λεπτό να βρω το χαρτάκι, η ανακοίνωση αφορά την, ότι η επικοινωνία συγγνώμη αφορά τα κράτη-μέλη, δηλαδή αρμοδία των κρατών μελών και το τι λένε τα κράτη-μέλη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά είναι ουσιώδε, είναι ουσιαστικό. Ε, πρόκειται για το σημείο 22-23, αν θυμάμαι καλά, για την ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Έτο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κυρία Επίτροπε. Αλλά να σα ε, αναφέρω ένα γεγονό ε, το οποίο έζησα προσφάτως στην χώρα μου, συναντώντας τους υπεύθυνους της επικοινωνίας της γαλλικής κυβέρνησης, παραπονέθηκαν για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χορηγούσαν παρά μόνο 800.000 ευρώ για να επικοινωνεί τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ τη Ευρώπη, Δηλαδή η Ευρώπη δεν θεωρούσε ότι θα έπρεπε να κάνει τίποτα θέματα επικοινωνία πέραν των 800.000. Νομίζω ότι αυτό είναι συνδοματικό σχέση με το ότι διαπιστώνουμε όλοι μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, απλέν τα πράγματα φτάνει οι Βρυξέλλε. Όταν ε, δεν πάνε στραβά, τότε δεν είναι οι Βρυξέλλε, είναι τα Λοιπόν, μέχρι ότι δεν κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε, να επερπηδήσουμε αυτέ τι πρακτικέ, ε, δύσκολα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον τομέα τη ευρωπαϊκή ταγένεια. Επίση, διαπιστώνω στη Γαλλία, αλλά θεωρώ ότι ισχύει και για πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ότι τα ευρωπαϊκά ζητήματα παραμένουν ως μια διεθνής ε, συνισταμένη μεταξύ άλλων αυτό το βλέπουμε και με την οργάνωση πολλών δικτύων και λυπάμαι γι' αυτό διότι όπως είπε και ο συνάδελφός μας 60 με 80% των αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. Δεν με ικανοποιεί πάντα, αλλά είναι φορές που με ικανοποιεί κάτι τέτοιο. Τώρα, ο προπολογισμό για το ευρωπαϊκό έτος της Ταγένειας θα είναι πολύ σύντομη, Πρόεδρε είναι ο πιο αδύναμος προπολογισμό ε, των τελευταίων ετών. Θεωρώ ότι δεν δίνουμε ένα πολύ καλό μήνυμα γιατί με την σημασία της ηθαγένειας ότι και αν πράττουμε σε συνδυασμό με άλλα προγράμματα και ειδικά με το πρόγραμμα Ευρώπη των Πολιτών. Ωραία, σας ευχαριστώ και τώρα η κυρία Παλιαδέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και υπόσχομαι να σύντομη. Ε, να επενέσω καταρχήν ε, ε, την πρόθεση της ε, Επιτροπής να γυρίσει στο παρελθόν προκειμένου να βοηθήσει στην Ευρωπαϊκή Συνοχή ε, και να, και να δηλώσει πως βεβαίως μέσω της επικοινωνίας αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Από αυτή την άψη επενώ επίσης και το website που θα γίνει απλοϊκό, απλούστερο ε, ε, προκειμένου να βοηθηθεί ο Ευρωπαίος πολίτης να ασχοληθεί ή να παρέμβει στα δρόμενα της Ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών οργάνων και πολύ περισσότερο περιμένουμε ε, πολύ ενδιαφέρον την ε, γωνιά των παιδιών, the kids corner όπως το ονομάσατε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από αυτές τις ηλικίε. Έχω μία ερώτηση μόνο. Ε, πραγματικά ο, η δημοσιογραφία είναι μεγάλο εργαλείο. Ε, θεωρώ ωστόσο ότι ο τρόπος με τον οποίο συχνά μεταφέρονται οι ερωτήσεις, οι, τα, γεγονότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαστρεβλώνονται και επηρεάζουν αρνητικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Ε, στην προσπάθεια λοιπόν της Επιτροπής και βεβαίως του ε, Κοινοβουλίου να φέρουν πιο κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες εκτιμάται πως θα μπορούσε να συμβάλλει ε, πέρα από τα σεμινάρια και μια μεγαλύτερη συνοχή σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρουπέλ, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Στην αρχή της ομιλίας σας είπατε ότι ο λόγος ύπαρξης της Ευρώπης είναι να ενδυναμώσουν τους πολίτες και οι πολίτες δεν γνωρίζουν συχνά τα δικαιώματά τους. Δυστυχώς αυτό είναι γεγονός. Και είπατε σωστά ότι η επικοινωνία θα πρέπει να, την επικοινωνία θα πρέπει να ακολουθεί και ένα μήνυμα. Αλλά ποιο είναι το μήνυμα διότι δεν μου κατέστη σαφές Τώρα πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, μπορούσε να, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι ζωτική σημασία. Οτιδήποτε φυσικά αν κάνουμε τώρα αφορά στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον του ευρώ. Και φυσικά ε, αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της ε, δικαιοσύνης. Αυτά, όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην στρατηγική της επικοινωνίας ε, που θέλετε να προωθήσετε. Thank you very much. It was just what I Ευχαριστώ. Και εγώ το ίδιο θα ήθελα να ρωτήσω. Πώς θέλετε να επικοινωνήσετε το μήνυμά σας. Ωραία, τελειώσαμε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Επίτροπη, διότι πρέπει να αναχωρήσει. Ο κύριος Γιούγκαργάρη δεν είναι εδώ λόγω του τέκνου του. Τι έγινε. Απέκτησε παιδί. Όχι, όχι, μιλάμε για πολιτικό τέκνο. Πολιτικό τέκνο. Ήθελα να το πω με ωραία και διαφορετικά λόγια. Έστω υπάρχει και αυτό το πάγωμα στον προπολογισμό. τώρα εσείς μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα. Παρακαλώ. Πριν απαντήσω συγκεκριμένα στα ερωτήματα των βουλευτών, κατάλαβα ότι η μνήμη και το μήνυμα προς, τους νέους, προς τις νέες γενιές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για χρηματικά θέματα, για χρηματοδότηση, για οικονομίες πρέπει να μιλούμε και για αξίες και για την κοινωνία. Μπορώ να σας πω από τη δική μου εμπειρία ότι αν επιμένετε οι πολίτες μονίμως άσχημα νέα ακούνε και πάντα χαίρονται να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι του δικού μας προγράμματος είναι αυτό που μπορούμε να μοιραστούμε. Έχω δει τις ε, αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πήγαμε από την Κεντρική Ευρώπη και προς το Βορρά και μετά προς την Ανατολή. Γιατί για μας ο φασισμός ήταν ε, πολύ ψηλά στην ατζέντα και μετά μπήκε και ο κομμουνισμός και τα πολιτερχικά καθεστώτα στην ατζέντα. Θέλαμε λοιπόν αυτό το κομμάτι της ιστορίας να το καταγράψουμε. Αυτό που δεν θέλω να γίνει, και νομίζω ότι και εσείς το ίδιο δεν θέλετε, είναι να μην υπάρξει ε, διαχωρισμός. Ότι να εδώ υπάρχουν ε, κάποιες ε, πράξεις που έγιναν παλαιότερα και ναι, αλλά είχαν γίνει και, και χειρότερα από κάποιους άλλους. Οτιδήποτε συμβαίνει κατά της ανθρωπότητας είναι of ε, φρικαλαιότητα. Η αναγκαιότητα να διατηρηθεί λοιπόν αυτή η μνήμη είναι μεγάλη. Εγώ έχω έρθει σε επαφή με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης για να δούμε και τα αποδερχεία καθεστώτα των ανατολικών χωρών και να μπει και αυτό στο όλο πρόγραμμα για το τι γίνεται με τη μνήμη και το τι θυμόμαστε. Ε, έχει προσθεθεί λοιπόν αυτό. Η δική σας ιδέα να υπάρξει ένα μουσείο για την κοινή μας ευρωπαϊκή ιστορία είναι Κάτι που ξέρω ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου το συζητούν για το πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Αλλά είναι σαφές ότι τα μικρά παιδιά και οι νέοι πρέπει να καταλάβουν τι είναι αυτό που ονομάζουμε πάνθεον και τι κάνουν τελικά, τι έχουν κάνει θετικό οι άνθρωποι. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε. Και χαίρομαι που ξεκινήσατε με την αναφορά στον Βάτσλαφ ε, Χάβελ. Είναι κάτι που μπορεί όντως να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των ε, νέων ανθρώπων. Το Euronews είναι ένα από τα εργαλεία επικοινωνίας που έχουμε. Σίγουρα δεν είναι το μόνο αλλά είναι ένα που πιστεύω ότι έπρεπε να διατηρηθεί και να διευρυνθεί, να του δοθούν περισσότερες γλώσσες ε, μετάδοσης. Ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Είναι όμως το μόνο που είναι όντως πολύγλωσσο και ευρωπαϊκό. Δεν έχουμε άλλο παρόμοιο. Γι' αυτό ήταν σημαντικό να παραμείνει, να παραμείνει ανεξάρτητο γιατί δεν μπορούμε να έχουμε εργαλείο επικοινωνίας που δεν είναι ανεξάρτητο. Και έπρεπε λοιπόν να το καταστήσουμε πιο γνωστό και να προχωρήσει την, ε, το έργο του. Θα οργανώσουμε λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, την ε, ε, επίσκεψη αυτή στα γραφεία του Euronews εδώ στις Βρυξέλλες και μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε μέσω του καναλιού αυτού. Συμφωνώ επίσης με την κυρία Χάνιβαλ. Η ενημέρωση είναι ακόμα κάτι τοπικό και ίσως να είναι και εθνικό. Γιατί αν δείτε το, τους αριθμούς των ανθρώπων που διαβάζουν εθνικές εφημερίδες ή αυτών που διαβάζουν τοπικές εφημερίδες, ο αριθμός των αναγνωστών τοπικών ε, εφημερίδων είναι πολύ μεγαλύτερος. Πολλές από τις πληροφορίες που παίρνουν είναι για τον τόπο τους και ε, έτσι καταλαβαίνουν καλύτερα τι γίνεται και αυτός ίσως να είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους δώσουμε αυτές τις ε, πληροφορίες. Να έχουμε δηλαδή τους κατάλληλους ε, δημοσιογράφους, οι οποίοι θα γνωρίζουν τον κάθε τόπο. Και πρέπει να έχουμε γι' αυτό κατάλληλη εκπαίδευση, για να τους δώσουμε τα εργαλεία, έτσι ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να κατανοήσουν πώς λειτουργούμε και εμείς εδώ, στα θεσμικά όργανα, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, τι γίνεται με τη συναπόφαση, πώς μέσω των ε, ευρωβουλευτών οι πολίτες μπορούν να παρουσιάσουν το σκεπτικό τους και να το μετατρέψουν σε απόφαση. Η κατάρτιση λοιπόν των δημοσιογράφων είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό το έχουμε τονίσει. Έχουμε τονίσει και τα σεμινάρια για τους για, να, για τους δημοσιογράφους, όχι για να τους ε, παρουσιάσουμε κάποιο δόγμα ότι εμείς είμαστε πολύ καλοί και κάνουμε την τέλεια, τέλεια δουλειά, αλλά για να, τους, ε, να δούνε πώς ακριβώς γίνεται η πραγματική ανάλυση, γιατί πολλοί λένε ότι δεν έχουν ε, το μέσο να κατανοήσουν το τι συμβαίνει. Ποιο είναι τώρα το μήνυμα που πρέπει να περάσει και γιατί δεν έχει μπει στο πρόγραμμα αυτό το μήνυμα. Γιατί το, πρόγραμμα δεν έχει να κάνει με ένα μήνυμα που ξεκινάει από πάνω και πάει κάτω. Το πρόγραμμα έχει να κάνει με την παροχή των εργαλείων ώστε να μπορεί να περάσει το, ε, μήνυμα. Το δικό σας μήνυμα, κυρία Χάνιμπαλ, και το δικό μου μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά τελικά είναι, είναι τα ίδια γιατί προσπαθούν να εξηγήσουν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα κεντρικό μήνυμα που θα περνάει προς τα έξω. Το, μόνο τα εργαλεία μπορούμε να διαθέσουμε στο, στην Κομισιόν, στο Κοινοβούλιο, στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, έτσι ώστε αυτά με τη σειρά τους να μπορέσουν να ενημερώσουν. Και μετά οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που θα περάσουν το μήνυμα στην κοινή γνώμη. Εμείς μόνο τα εργαλεία μπορούμε να τους δώσουμε, ώστε η κοινωνία των πολιτών να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα για να γίνουν ας πούμε οι αδερφοποίησεις των πόλεων, για να μπορέσουν να γίνουν συναντήσεις των νέων ή οτιδήποτε άλλο. Και το ίδιο έχει να κάνει με, την, ε, με το Ευρωπαϊκό Έτος όχι της Ιθαγένειας, αλλά των πολιτών. Το κατέστησα απόλυτα σαφές. Είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των πολιτών. Και δεν είναι το θέμα μας μόνο το ελεύθερη διακίνηση, γιατί είδαμε και το θέμα του οδικού χάρτη και πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ελεύθερης διακίνησης. Και θέλω να σας πω ότι υπήρξαν 16 κράτη-μέλη όχι μόνο η Γαλλία, που έπρεπε να αναθεωρήσουν τα εθνικά τους προγράμματα, γιατί δεν είχαν προσαρμόσει την ε, οδηγία πλαίσιο του 2004. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξηγήσουμε στους πολίτες ποια είναι τα δικαιώματά τους, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης και ποιες είναι οι ευκαιρίες τους. Αν δείτε δηλαδή τους φοιτητές, αν δείτε τους επαγγελματίε. Νομίζω ότι εδώ όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να ε, και να πάνε κοντά στους πολίτες αυτά, στα πλαίσια αυτού του έτους. Ε, δεν χρειάζεται να βρούμε έμιστους για να κάνουν αυτό. Το, το πράγμα πρέπει να, να, να εμείς να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε και να βγούμε στους πολίτες και να τους μιλήσουμε. Οπότε πάω σε κάποιο εθνικό κοινοβούλιο ε, Συγγνώμη τώρα που μιλώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εθνικά, αλλά όποτε μιλώ για το, ε, εθνικό, για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, τους λέω ότι αυτό το έτος είναι δικό σας. Όταν πάω στην Επιτροπή των Περιφερειών, μιλάω με τον, με τον Πρόεδρο, με τα μέλη και τους λέω ότι είναι δικό σας αυτό το έτος. Και ο καθένας πρέπει να λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να πάει στους πολίτες και να εξηγήσει τι ακριβώς κάνουμε στην Ευρώπη για τους πολίτες. το κόστος αυτού είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αισθάνομαι πολύ περήφανη για το πρόγραμμα των πολιτών που έχει παραμείνει στον προϋπολογισμό και δεν έχει μειωθεί. Είναι 30 εκατομμύρια ή λίγο παραπάνω, δεν είναι κακό. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα το περικόψει, κυρία Πρόεδρε, την επικοινωνία. Είμαι, δεν είμαι από αυτούς που καταβροχθίζουν τα κονδύλια και πραγματικά πρέπει να συνεργαστούμε για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λίγα χρήματα. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δείξουμε στους πολίτες ότι δεν είναι τα χρήμα μόνο αυτό που μετράει, αλλά είναι οι άνθρωποι. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ελευθερίες, με ρίζες και η νέα στιγμή της Λισαβόνας ε, μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε με Ευρώπη των δικαιωμάτων, Ευρώπη της δικαιοσύνης. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη χρονιά προκειμένου να το πετύχουμε. Και κυρία Βεζιά, θα πρέπει να βάλουμε μέσα αυτά που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητα και σημαντικά. Εγώ όταν πηγαίνω στους Λουξεμβουριανούς πολίτες ε, μιλάω με ένα διαφορετικό τρόπο παρά όταν πηγαίνετε εσείς παρά ε, μάλλον και εσείς μιλάτε διαφορετικά όταν απευθύνεστε στους πολίτες σας, στη χώρα σας, στη Γαλλία. Έχουμε πρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος ευτυχώς μιλάει για τα καλά που κάνει η Ευρώπη για την χώρα του. Το σημείο κίνηση λοιπόν το δικό μου είναι ευκολότερο. Αλλά δεν πάω μόνο στο Λουξεμβούργο, πηγαίνω και στη Γερμανία, πηγαίνω συχνά στην χώρα αυτή. Και εκεί πρέπει να προσαρμόσω το μήνυμά μου, χωρίς όμως να αλλάζω την ουσία του μήνυματος. Η ουσία παραμένει ίδια, αλλά μιλάω διαφορετικά στους Βαβαρούς και διαφορετικά στους ε, πρώην Ανατολικογερμανούς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς που φέρουμε ευθύνη ε, θα πρέπει να προωθούμε το μήνυμα με τον καταλληλότερο των τρόπων ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Η γωνιά των παιδιών τώρα. Πρέπει να τη δούμε για να καταλάβουμε είναι, αν είναι το σωστό εργαλείο που χρειαζόμαστε, αν θα πρέπει να το οργανώσουμε με διαφορετικό τρόπο. Και επί τη ευκαιρία. Και τα παιδιά είναι πολίτες. Πρέπει να έχουν το χώρο τους στη διάρκεια του, του ευρωπαϊκού έτους υπηκότητας. Και ευτυχώς έχουμε εξαιρετικούς δασκάλους, όχι, όχι αρκετούς. Και δυστυχώς έχω διατελέσει επίτροπος παιδείας και γνωρίζω ότι οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τα σχολεία είναι μηδέν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προτείνουμε, να παράσχουμε τα μέσα στους δασκάλους και οι δάσκαλοι να τα χρησιμοποιήσουν, να προσφέρουν τις ευκαιρίες στα παιδιά μέσω αυτής της γωνίας των παιδιών στο διαδίκτυο, να τα προσελκύσουμε ίσως. Θα έρθουν σε επαφή μαζί σας. Δεν είναι θέμα της Κομισιόν να επικοινωνήσει. Η κυρία Πρόεδρος ρώτησε σχετικά με το τηλεοπτικό δίκτυο. Ξέρω ότι αυτό είναι το δικό σας παιδάκι, της Επιτροπής σας του κύριου Λόκογκαρτ, αλλά ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής σας και υπήρξε εισηγητής. Και εσείς το επιθυμούσατε. Είναι καλή ιδέα, θεωρητικά. Αποδείχτηκε μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες που φτιάξαμε, μια διαδικασία καταρχήν προμηθειών το 2008-2010, όπου επιλέξαμε υποψηφίους, είχαμε διμερή διάλογο, διαδικασίες δημοπράτησης και μετά την αξιολόγηση των προσφορών του 2010, μια ενδελεχή ανάλυση που έκανε ομάδα ανεξάρτων εμπειρογνωμόνων από την Κομισιόν αλλά και από το Ευρωπαϊκό Τηλεοπτικό Παρατηρητήριο. Στο, συμμετείχε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με έναν παρατηρητή σε μία ομάδα. Τρεις προτάσεις έφτασαν στην τελική φάση. Η μία παρέμεινε. Και δεν ναι, μία δεν ανταποκρίθηκε στην ε, καλή ιδέα που είχε αρχικά το Κοινοβούλιο. Και έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει κανείς να το ξανασκεφτεί. Με τους ελάχιστους πόρους που διαθέτουμε. Αξίζει το κόπο να επενδύσουμε σε κάτι που θεωρούμε ότι δεν θα πάρει μπρος. Όπου ο κίνδυνος είναι ψηλός αλλά τα λεφτά πολλά. Μιλάμε τώρα για 8,3 ε, εκατομμύρια ευρώ τις πρώτες χρονιές και 10 τις τελευταίες. Αν το συγκρίνετε με τα 228 εκατομμύρια που έχουμε στον προπολογισμό για τους πολίτες, αντιλαμβάνεστε ότι για μας πρόκειται για μεγάλο ποσό. Οπότε, θεώρησα ότι όχι, δεν θα ήταν σωστό να δαπανηθούν έτσι τα χρήματα, όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες. Εσείς κυρία Πρόεδρε λάβατε επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία μπορείτε να κοινοποιήσετε στους συναδέλφους. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε σχετικά. Όλα εξελίχθηκαν σύμφωνα με την, ε, έγιναν κατά τον πρέποντα τρόπο. Τα χρήματα λοιπόν τι έγιναν. Όχι, δεν πήγε μόνο στο Euronews. Το Euronews πήρε μέρος του κοντιλίου αυτού. Το δώσαμε στο SCAD Plus. τις ε, ανακεφαλαιώσεις ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στις 22 επίσημες γλώσσες. Και εσείς στην Επιτροπή σας το είχατε σκεφτεί, είχε... πήγαινε για κατάργηση. Πήρα λοιπόν ένα μέρος του κονδυλίου για να το βάλω στην ιστοσελίδα και ένα μέρος στα Euronews. Καταναμήθηκαν λοιπόν αυτά τα χρήματα και συμφωνώ ότι θα πρέπει ίσως και αργότερα να συζητήσουμε. Έχετε εδώ κάποιον που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα απτικοακουστικά, ο Γενικός Διευθυντής, ο Γκρέκορι Πόλτσε, θα είναι στη διάθεσή σας τον Ιανουάριο με μια, ένα πρόγραμμα ανακοίνωσης και θα δούμε μετά εάν υπάρχουν θέματα που θέλετε για να προωθηθούν τα μηνύματα με διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Μόνο μία πρόταση για αυτό το, την πανευρωπαϊκή συζήτηση. Εμείς την ψηφίσαμε, αρχίσατε κάτι να κάνετε, διαπιστώσατε ότι δεν λειτουργεί και μετά το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι να έρθετε να μας πείτε, ακούστε, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, η αξιολόγηση μου λέει ότι δεν αξίζει τον κόπο και έδωσα τα χρήματα εκεί και εκεί και εκεί. Έτσι το καταλαβαίνουμε καλύτερα και το χωνεύουμε καλύτερα. Το μάθαμε με άλλο τρόπο και ο κ. Λόκακάτ είχε εξοργιστεί, αλλά το καταλαβαίνουμε. Είμαστε στο τέλος του έτους. Πάντοτε κάνουμε, παίρνουμε τις αποφάσεις μας για το επόμενο έτος. Μάθαμε από αυτή την υπόθεση ήρθα στο τέλος της υπόθεσης αυτής, όχι στο ξεκίνημα, δεν ήμουν εδώ. Αναλαμβάνω όμως όλη την ευθύνη για το πώς ολοκληρώθηκε, πώς τελείωσε. Τώρα πια μπορώ να σας πω ότι αν υπάρξει άλλη τέτοια υπόθεση θα τη χειριστώ διαφορετικά, καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, διακόπτουμε για ένα δίλεπτο για να ξαναρχίσει Je te donne la parole pour, euh, pour présenter ton draft. Λοιπόν, πολλά είπε, προηγουμένω, γι' αυτό α ε, συντμήσει λίγο τα όχι. Μπορώ να ακούσω και του υπόλοιπου αν θέλει. δεν έχω λόγο να, ε, πάρω, να μιλήσω. Καταρχήν λοιπόν, να πω ότι λυπάμαι για τους ε, περιορισμούς με τις ημερομηνίε. Τη στιγμή που το σχέδιο χρωμοδότησης, που είμαι υποχρεωμένη να στείλω το σχέδιο χρωμοδότησης για μετάφραση, έχει φτάσει και δεν μπορώ λοιπόν να λάβω υπόψη μου τις παρατηρήσεις που γίνονται. Λαμβανωμένο αυτού υπόψη συνεργάστηκα με τους Σκιώδης εκ των προτέρων και συνεδριάσαμε δύο φορές για να προσπαθήσουμε κάτι να κάνουμε ε, που να συγκλίνουν, στο οποίο να συγκλίνουν οι απόψεις. Δεν έχουμε ε, μεγάλες διαφορές διαφωνίες μεταξύ μας. Η ουσία είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως Νομίζω ότι όλοι εδώ συμφωνούμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ή μάλλον ότι ε, στο θέμα της υπηκότητας δεν βλέπουμε μόνο το δικαίωμα ψήφου, το στο δικαίωμα, αλλά και την ε, εκπαιδευτική και πολιτιστική διάσταση της ηθαγένειας. Προσπάθησα αυτό να το βάζω με τη μορφή τροπολογίας την γνωμοδότηση αυτή λαμβάνοντας υπόψη όλο το, όλες τις ε, θεσμικές διατάξεις που έχουμε και όχι μόνο τα άρθρα 20 και 21 της συνθήκης και κάνοντας κάποιες προτάσεις ε, σε κάποια θέματα, ας πούμε για την παιδεία, τον πολιτισμό, την κινητικότητα των φυτών. Θα απαντήσω και σε ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο κ. Ρίκγκαρτ που είναι σκιώδης μαζί μου έχει υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες που θα λάβουν καλύτερα υπόψη τα στοιχεία της έκθεσης που αφορούν την επικοινωνία γιατί είναι πιο ειδικός από μένα στα θέματα αυτά. Το άλλο στοιχείο, η άλλη διάσταση που έλεγα προηγουμένως είναι ότι μάλλον πρέπει να στηρίξουμε τις, υπόψη, τις προσπάθειες της Επιτρόπου ε, για να ξεκινήσει εκ των κάτω η όλη αυτή η προσπάθεια και όχι εκ των άνω. Ε, υπάρχει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να υπάρξουν παντού. Εγώ αποδίδω ιδιαίτερη, εντελώς ιδιαίτερη σημασία στο να ληφθούν υπόψη η κοινωνία των πολιτών και οι εκπρόσωποι τη, έχοντας πάντοτε κατά νου το πολιτιστικό τομέα που διαθέτει πιστεύω δίκτυα τα οποία μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα συμπεριλαμβανομένης και αυτής της περιπτώσεως. Ε, κάτι άλλο που επίσης δεν με ευχαριστεί λόγω της ε, ειδική ε, φύσης της έκθεσης αυτής που είναι νομοθετικού περιεχομένου υπάρχουν ακόμα μεγαλύτεροι περιορισμοί δεν ήταν εύκολο γιατί εγώ πρέπει να πω ότι δεν έχω αναλάβει άλλη έκθεση οπότε δεν είναι όλα τα πράγματα πολύ απλά. Θα ήθελα, όπως έλεγα και πριν, να συμπεριλάβω στην πρώτη αυτή πρόταση μια τροπολογία για την δημοσιονομική διάσταση την οποία, ε, η οποία μου είναι ιδιαίτερος ε, προσφυλής. Αναφέρομαι στο ότι αυτή τη στιγμή το σχέδιο έφυγε χωρίς αυτό. Λυπάμαι γιατί ε, ε, έφυγε όπως την εξέταση η νομική υπηρεσία. Θα ήθελα λοιπόν να ληφθεί υπόψη αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ πολύ περίεργο ένας... Ε, να μην αναφέρεται στο θέμα αυτό της ηθαγένειας, αυτό ο περιορισμένος προϋπολογισμός των τελευταίων ετών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Ο κύριος Μπόγονς. Ε, Ευχαριστώ. Να ζητήσω από την εισηγήτρια να μου πει αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εξέλιξη των ε, κρατών μελών, όχι μόνο την κοινοτική πτυχή. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις ε, περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και τις διάφορες οργανώσεις. Εσείς θα υποβάλλετε τέτοιες, θα κάνετε κάποιες τέτοιες αλλαγές στο κείμενο ώστε να ενισχυθεί αυτό το μήνυμα, το οποίο έχει στόχο τα κράτη-μέλη, την Επιτροπή των Περιφερειών, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών να γίνει μια κοινή προσπάθεια ένα κοινό εγχείρημα, γιατί μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδες μεμονωμένων ε, δραστηριοτήτων σε, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ, κυρία Στεναλόγα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τα πω καλά στα αγγλικά. Να ευχαριστήσω την κυρία Βερζιά για την πολύ καλή συνεργασία με τους σκιώδεις συζητητές. Κάναμε πολλές συναντήσεις και Η έκθεση έχει όντως πάρα πολλές ε, πτυχές. Τις ε, συζητήσαμε και πριν από λίγο με την Επίτροπο Ρέντινγκ, γιατί μιλούμε και για την ευαισθητοποίηση για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, για την επικοινωνία, για τη συμμετοχή, Βεβαίω, ε, και οι συνθήκες και η χάρτα ε, εξασφαλίζουν ε, την συμμετοχή και την πρόσβαση των πολιτών σε όλα αυτά τα έγγραφα στη γλώσσα τους και να μπορεί κανείς να λάβει ερώτηση στο στο, απάντηση στο ερώτημα που θέτει. Οι περισσότερε όμω διαβουλεύσει συνήθω γίνονται μόνο στα αγγλικά ή ίσω και στα γερμανικά και γαλλικά. Αν λοιπόν θέλουμε όντω του ευρωπαίου πολίτε να συμμετέχουν και να μπορούν να εκφράσουν την άποψή του σε αυτές τις δημόσιες διαβουλεύσεις και να συμμετέχουν πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα μπορούν να γίνονται σε όλε τι επίσημε γλώσσε. Και πρέπει επίση να καταστήσουμε το σύστημα το όσο δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη γίνεται. Επίσης, ως κοιόδη συγγήτρια για αυτή την πρωτοβουλία, πρέπει να πω ότι πρέπει να τονίσουμε και τη σημασία αυτού του εργαλείου. Και τέλος, να δούμε και την διανομή των πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο και την ενημέρωση των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών και οργανώσεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντική και η πολιτιστική πτυχή του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών. Μιλούμε για την ε, μάθηση και την ε, αναγνώριση όλων των ε, πολιτισμών και των κοινών μας αξιών. Όταν εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγώ Κάθε έξι μήνες στην πόλη μου ξεκίνησα να οργανώνω ε, ημέρες πολιτισμού για την ε, χώρα για την οποία ανέλαμβανε την, ε, την ε, Προεδρία του Συμβουλίου πριν από λίγο ολοκληρώσαμε, πριν από λίγες μέρες ολοκληρώσαμε την ε, παρουσίαση για την Πολωνική Προεδρία. Κάθε φορά το, η εκδήλωση αυτή έχει όλο και περισσότερους υποστηριχτές, όλο και περισσότερους ε, προσεκλημένους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες. Όσο πιο κοντά είμαστε τόσο καλύτερα. Γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε μεγάλη συνδιάσκεψη. οι 754 ε, ευρωβουλευτές δεν θα μπορούσαν να οργανώσουν κάτι παρόμοιο για τους πολίτες τους. Ε, ίσως να είναι πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Βερζιά για την ε, προσέγγιση που έλαβε σε σχέση με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Elnök asszony, θα είμαι σύντομος αυτή τη φορά. Μιλούμε για την ε, πολιτισμική και θρησκευτική πτυχή. Σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά θέματα, μιλούμε για το διάλογο μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Έτος, Νομίζω ήταν το 2008 το έτος αυτό, το ευρωπαϊκό έτος και ήταν πολύ επιτυχές το έτος του πολιτισμικού διαλόγου. Ο πολιτισμός φέρνει κοντά τους πολίτες, καθώς επίσης και η, α, η θρησκεία. Στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου εγώ είμαι υπεύθυνο για τον διάλογο με τις ε, εκκλησίες. Ε, σημείο 17 στη συνθήκη της Εκεί υπάρχει διάταξη που μιλάει για τις εκκλησίες ε, οι οποίες είναι καθολικοί οργανισμοί και είναι μια πολύ καλή βάση ε, όπου μπορούν να έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι μέσω της πίστης. Γι' αυτό οι εκκλησίες μπορούν να παίξουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το έτος των πολιτών. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Να ε, καθησυχάσω το συνάδελφο για τα διάφορα ε, επίπεδα εμπλοκής που αναφέρομαι στην έκθεση. Κάθε φορά που είναι δυνατόν, νομίζω τουλάχιστον εγώ, όχι μόνο έχουμε προσπαθήσει να στείλουμε μήνυμα προς τους εμπλεκόμενους από την κοινωνία των πολιτών αλλά και στις δημόσιες αρχές οποιοδήποτε επίπεδο γιατί θεωρώ ότι η ηθαγένεια ζει σε κάθε επίπεδο και δεν μπορούμε να την ε, βάλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν δεν λειτουργεί στο χαμηλότερο δυνατό, στο πεδίο και πιστεύω ότι οι τοπικοί άρχοντες είναι σημαντικοί, Αδερφοποίηση είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα όσο περισσότερο ενισχύονται, συμπεριλαμβανομένων και στον εκπαιδευτικό τομέα θα καταφέρουμε να ζήσει αυτή η ευρωπαϊκή ηθαγένεια σε όλες τι τις διαστάσεις. Το γλωσσικό ζήτημα προσπαθήσαμε να το δουλέψουμε αρκετά. Ε, είναι σημαντικό, έχουμε να κάνουμε πραγματική μάχη, γιατί αν δεν καταφέρουμε να ενημερώσουμε τους πολίτε τη γλώσσα τους, τότε ε, θα δεν θα υπάρχει συνεννόηση. Όσον αφορά τα θρησκευτικά θέματα δεν επισέρχομαι σε αυτά γιατί θεωρώ ότι μάλλον διαιρέσεις και όχι ενότητα θα προκαλέσω. Προσπάθησα λοιπόν στις ε, τροπολογίες που προτείνω να, είναι, να κινηθώ συνενετικά ώστε να μπορέσουμε όλοι να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση ώστε η ευρωπαϊκή θαγένεια να επιτύχει. Επανέρχομαι και πάλι στο δημοσιονομικό ζήτημα κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπάρξει κυρία Πρόεδρε Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πραγματικά στην τροπολογία που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει και δημοσιονομικό ε, τροπολογία. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Θα ήθελα να έχω τη συνεργασία των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Να κλείσουμε το θέμα. Οπότε ερχόμαστε Εξυγχρονίζεται τώρα το, Ευρωπαϊ... το... Κύριε στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη. Uh, Είναι η πρώτη μου έκθεση Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη έκθεση στην Επιτροπή αυτή. Αφορά τον εξυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων είχε προγραμματιστεί για στις 23 Νοεμβρίου. Τελικά, με μεγάλη χαρά, στην, ε, μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού, να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 19 εκατομμύρια μυθητές και πάνω από 500 ε, ε, ιδρύματα φάσμα εκπαίδευσης και παρότι θα το 35% όλων των θέσεων εργασίας του 2020 θα απαιτεί εξειδικευμένη εργασία. Αυτή τη στιγμή μόνο το 26% του εργατικού δυναμικού έχει ε, προσόντα υψηλού επίπεδου. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη για εξυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Η έκθεσή μου αυτό αφορά Η έκθεση θα παρουσιάζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Η ευθύνη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται κυρίως στο επίπεδο των κρατών μελών και στα ίδια τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα προγράμματα Εράσμους συμπληρώνουν και συντονίζουν τις προσπάθειες των κρατών μελών. Κατά την ε, σύνταξη του σχεδίου έκθεσης, θέλω να ευχαριστήσω την Μιχαήλα Φάιφερ, της γραμματείας του, της, ομα, του, της ομάδας, τον Ρομπέρτο Τιζενέλα, τον Κούρτ και τον κύριο Άνταμ Τάισεν από το ΕΛΚ, με τους οποίους διαβουλεύτηκα. Και τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την σύνταξη της ανακοίνωσης. για την ευκαιρία να διαβουλευτώ με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, τον κύριο Μάικλ Γκέιμπλ, επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής και, εκπρόσωπο, και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, φοιτητών, την πρόεδρο Καρίνα Ούφερτ. Επίσης ε, συναντήθηκα με τους υπεύθυνους στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι Ο περιορισμένος αριθμών λέξεων που πρέπει να έχει η έκθεση της πρώτη, του το πρώτο σχέδιο έκθεσης περιορίζει θέματα που μπορεί να συμπεριληφθούν, όπως επίσης και την παρουσίαση κάποιων θεμάτων. Όμως η περαιτέρω διαδικασία θα μας επιτρέψει να εισάγουμε στην έκθεση περαιτέρω στοιχεία ή να ε, αναφερθούμε λεπτομερέστερα σε αυτά που ήδη θέτουμε. Επικεντρωνόμαστε σε βασικά σημεία του σχεδίου έκθεσης, τα οποία είναι τα εξής. Η ενίσχυση και η προώθηση των ε, τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συνεργασία με όλους τους εξωτερικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένων και των, ε, του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και τα ε, συμβούλια δημόσιας διοίκησης, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και την ευρύτερη κοινότητα της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη για εξωτερικούς εταίρους οι οποίοι θα πρέπει να ε, συμμετέχουν σε αυτή τη συνεργασία δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες ε, περιφερειακές αλλαγές, ε, διαφορές στα κράτη-μέλη στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα άλλο θέμα που είναι κεντρικό είναι η ανάγκη για μεταρρύθμιση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν μεγάλες αλλαγές ε, στους φοιτητές τους, δηλαδή ενήλικες ε, ε, επαγγελματίες και μη παραδοσιακούς φοιτητές. Χρειάζεται που χρειάζονται να αναβαθμίσουν ή να αναδιαμορφώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Χρειάζεται στενή συσχέτιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας η ενίσχυση της μετάβασης από το ένα είδος ε, ιδρύματος σε άλλο, από το ένα επίπεδο στο άλλο, από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Η υποστήριξη των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συμμαχίες γνώσεων, τις ε, συμμαχίες των ε, διαφόρων τομέων, την ανάγκη για αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία για την διαδικασία εξυγχρονισμού και επίσης ένας μεγαλύτερος προπολογισμό για την παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να συνεργαστεί με χώρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες να συμπεριληφθούν όλες οι κοινωνικές, εθνικές και υπο ε, αντιπροσωπευόμενες ομάδες. Θα πρέπει η τριτοβάθμια εκπαίδευση να θεωρείται ένα δημόσιο αγαθό που ενισχύει την πολιτιστική πολυπλοκό, ε, ε, πολυμορφία και την ενεργό ε, συμμετοχή των πολιτών. Τέλος, θέλω να επισημάνω δύο στοιχεία. Πρώτον, τις διαφορές που υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επειδή προέρχομαι από την Ανατολική Ευρώπη, μπορώ να επιβεβαιώσω το ότι εμείς έχουμε μείνει πίσω. Από τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, μόνο 200 ε, βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτά τα 200 κανένα ή ίσως πολύ λίγα ε, βρίσκονται σε χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η ενσωμάτωση λοιπόν, η ολοκλήρωση θα πρέπει να συμπεριλάβει και τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι πρέπει να προσφέρεται τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μειονοτικές γλώσσες. Εμείς είμαστε Ουγγροί από τη Ρουμανία και έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Για μας η Βέλγη είναι παραδείγματο χάρη η τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχει η Φιλανδία, όπου η, η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη σουηδική γλώσσα είναι ισοδύναμη με αυτή που παρέχεται στη φιλανδική γλώσσα. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί και να εξυγχρονιστεί το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, όσον αφορά τη σύνταξη, και επειδή ε, έχουν τεθεί όρια, θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ζητήσω να υποβάλλετε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό τροπολογιών, γιατί εκεί δεν έχουν δεν υπάρχουν όρια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τόκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση της έκθεσης. Τους προηγούμενους μήνες ε, μιλήσαμε πολλές φορές για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη σε σχέση και με την έκθεση πρωτοβουλίας ε, του Berlinguer και δεν έχω να προσθέσω πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ώστε η έκθεση που έχουμε εδώ για την ανακοίνωση να είναι συνεπής και συνεκτική με την έκθεση πρωτοβουλίας. Έτσι ώστε να είναι συνδεδεμένες οι δύο αυτές οι εκθέσεις μεταξύ τους και να έχουμε συνολικό, μια συνολική πρόταση η οποία θα κινείται προς σωστή κατεύθυνση να μην ε, έχουμε δηλαδή, να κάνουμε δύο φορές την ίδια δουλειά, πρώτα για την ε, ε, ανακοίνωση και μετά για την έκθεση πρωτοβουλίας, να μην υπάρχουν αντιφάσεις, να έχουμε λοιπόν ένα καλό κοινό σύστημα. Και ειδικά σε ό,τι αφορά το Εράσμος, Έχουμε και την, έκθεση, την πρόταση συγγνώμη της Κομισιόν για την χρηματοδότηση των ε, προεκπαιδευτικών προγραμμάτων και σε αυτό το τομέα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και κατά πόσο τα διάφορα αιτήματα που υπάρχουν για, τον, ε, για το Εράσμος για τη νέα πρόταση τέλο πάντων για όλα τα προγράμματα, αν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σε ό,τι αφορά την ε, ε πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ας πούμε, αν έχω καταλάβει καλά, στο μέλλον θα υπάρξουν ε, για τους φοιτητές μάστερ ε, κονδύλια από το Ταμείο Εγγύσεων, αλλά στο μέλλον δεν θα δίνεται υποτροφία Εράσμους στους φοιτητέ Εράσμους. Αν έχω καταλάβει καλά, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ προβληματικό. Οι περισσότεροι φοιτητέ συνήθω πάνε στο εξωτερικό για το μάστερ του. Εκτό αν δεν έχω καταλάβει εγώ. Αλλά τουλάχιστον εγώ έτσι διάβασα την πρόταση τη Κομισιόν μέχρι στιγμή. Ότι δηλαδή θα υπάρχουν για του ε, φοιτητέ μάστερ ε, κονδύλια μόνο από το Ταμείο Εγγυήσεων. Αν τώρα το πράγμα είναι έτσι, αυτό ας πούμε είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε εδώ να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση, αλλά ίσως πάλι λέω να έχω καταλάβει κάτι λάθος εγώ. Οπότε θα μπορούσαμε να το διευκρινίσουμε και να το ερευνήσουμε ε, καλύτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και πάλι λέω να τα συνδέσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις. Ο κύριος Μπόρης. Ja ogromnie się cieszę, że e, kolega Laszlo zajmuje się tym sprawozdaniem. E, Χαίρομαι που ο κύριος ε, Λασλοτόκης ασχολείται με την ε, έκθεση. Είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με το ζήτημα της ε, μη αναλογικότητας, δηλαδή το θέμα των πανεπιστημίων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Θα πολύ ευχαρίστω να συνεργαστούμε σε επίπεδο τροπολογιών, διότι όπως είπατε είναι περιορισμένη τυπικά η έκθεση ενώ οι τροπολογίε, για τι τροπολογίε δεν υπάρχει κανένα περιορισμό. Πρέπει να ασχοληθούμε με την. Ε, ε, με τη στρατηγική Ευρώπη του 2020 θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα ανώτερο ποσοστό αποφύτησης ε, των μαθητών από το σχολείο τώρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε επίση και στην ποιότητα της παιδείας. Ξέρουμε ότι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Η δημογραφία έχει αρχίσει να αλλάζει και στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Επίσης γνωρίζουμε ότι ενδεχομένω κάποια δημόσια πανεπιστήμια θα εξαφανιστούν και στη θέση τους θα εμφανιστούν ιδιωτικά. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι ότι ο κύριος Τόκες μίλησε για την προσαρμογή των πανεπιστημίων στις απαιτήσει ε, της αγοράς εργασίας. Αυτό είναι ζήτημα που τίθεται πανταχού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε 10-20 χρόνια δεν ε, θα κατορθώσουμε να προσαρμόσουμε τα φοιτητικά προγράμματα, προγράμματα στις ανάγκες αγορέ. Μερικέ φορέ υπάρχουν ελλείψεις ε, στο ρεμέ προφορικής. Έχουμε ελλείψεις σε ε, θέματα παροχής ε, νοσοκομειακών νοσοκομιακής περίθαλψης νοσηλευτριών και νοσηλευτών. Και αυτό θα και αυτό, αυτό πρέπει να μας οδηγήσει στο να δημιουργήσουμε προγράμματα συνεργασίας ε, με πολλά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα με αυτά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, διότι υπάρχει μια δυσαναλογία και αυτή θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Ευχαριστώ. Ξέρετε, θα είναι δύσκολο να καταρτήσει την έκθεση αυτή ε, δίχως ε, να υπάρξουν αντιφάσεις, ε, αλλά παρακαλώ να φροντίσετε να διορθώσετε κάπως την έκθεση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στο ζήτημα των μάστερ και της κινητικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει μια εγγύηση προς τις τράπεζες που θα χορηγούν δάνεια στους φοιτητές που θέλουν να ολοκληρώσουν το μάστερ τους. Πρόκειται λοιπόν για έναν, έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στις τράπεζες να αυξήσουν την παροχή δανείων σε φοιτητές. Θα υπάρξει ένα είδος μόχλευσης αν θέλετε και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η Κομισιόν προτείνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέχει τις εγγυήσεις ε, προκειμένου να λαμβάνουν δάνεια οι φοιτητές. Τώρα για την ανακοίνωση στο σύνολό της Αναφερθήκατε, ε, μάλλον η Επίτροπος αναφέρθηκε σε πέντε ζητήματα που αφορούν την ε, εκπαίδευση, ο αριθμός ε, των φοιτητών, ε, η ποιότητα της, ε, των σπουδών. Ο Μπορείς επίσης αναφέρθηκε στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κινητικότητα σε επίπεδο διασυνορικής συνεργασίας. Μέχρι τώρα το πρόγραμμα εράσμους είχε τεράστια επιτυχία, όπως και με το Βούντες και το Τέμπους, ε, Επίση υπάρχει το ζήτημα της αναγνώρισης ε, των προσόντων, ε, το οποίο εξετάζει η έκθεση Όταν όμως προσπαθούμε να πετύχουμε συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, Ξέρετε ότι αυτό καθίσταται μερικές φορές ιδιαίτερα δύσκολο και περίπλοκο σε κάποια κράτη. Και τέλος, το ζήτημα της χρηματοδότησης. Δεν θέλω να υψέρθω σε λεπτομέρειες εδώ. Αυτό που θα ήταν χρήσιμο είναι οι θέσεις του Κοινοβουλίου σε μια σειρά δράσεων αναφερθήκαμε σε ένα διάφανο σύστημα ε, βάσει το οποίο θα πρέπει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Ακούσαμε την ε, πρωτοβουλία για την κινητικότητα στο πλαίσιο του Εράσμους. Προσπαθούμε να προωθήσουμε στρατηγική συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων κάτι το θα οδηγήσει σε πιο διαρθρωμένη ανταλλαγή προσωπικού αλλά και φοιτητών. Και τέλος, πιο στρατηγική χρήση των ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σε ζητήματα κατάρτισης, αλλά και για τον ε, προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα, όλα αυτά θα μπορούσαν να συνδυαστούν για να αντιμετωπίσουν όλες τις πτυχές ε, του εξυγχρονισμού των συστημάτων της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τις θέσεις του Κοινοβουλίου πάνω στα ζήτημα. Θα υπάρχει το Erasmus for All, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματά του σχετικά με την ατζέντα περί εξυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης εκπαίδευση. Δέχτηκε πολλέ από τι προτάσει τη Κομισιόν και με μεγάλη ικανοποίηση θα δεχθούμε και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για το θέμα. Να επανέλθουμε λίγο στο ερώτημα που τέθηκε πριν. Γιατί είπε η συνάδελφος ότι για, το, για τα μάστερ. Για τα μάστερ είπαμε θα υπάρχουν δυνατότητες και από το βασικό πρόγραμμα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ήταν δυνατό για, για το σύνολο των σπουδών μάστερ να ε, χρηματοδοτηθεί. Δεν μιλάμε για το Εράσμους λάθο, ε, παρανόηση υπήρξε, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Ε, κάποτε δασκάλα ήμουνα, τι να κάνω, δεν μπορεί να μου φύγει το κουσούρι. Φαίνεται, ε. Λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Τάισον. Ο κύριος ε, και πάλι. Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε. képviselőtársammal Προτού να προετοιμάσω την τελική έκθεση, ε, συναντήθηκα και με τον κύριο Μπερλιγκουέρ, που είναι σκιώδης ηγητής επί της συγκεκριμένης εκθέσεως. Ε, Συζητήσαμε λοιπόν το θέμα και είμαι σε θέση να πω ότι τόσο η δική του έκθεση όσο και η δική μου έχουν το στοιχείο της που Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε και τις ε, επικαλύψεις. Σε ό,τι φορά το πρόγραμμα Erasmus και Erasmus Master Degree Mobility Scheme είναι δύο πρωτοβουλίες ε, ιδιαίτερα σημαντικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας. Και τώρα θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας ε, σε ένα θέμα. Η σχέση μεταξύ κινητικότητας και διαρροής ε, μυαλών. Εμείς ε, με ιδιαίτερη απογοήτευση βλέπουμε να εγκαταλείπουν την, τις χώρες μας ε, εγκέφαλοι Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά ε, εκπαίδευση ανώτερη φτερή της τριτοβάθμιας, δηλαδή δοκτορά ε, και περαιτέρω εξειδίκευση των πτυχιούχων. Υπάρχουν άλλες χώρες που ελκύουν αυτά τα, αυτούς εγκεφάλους και θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να ξεύρει μια λύση στο ζήτημα. Εντάξει, θα είναι δύσκολο το εγχείρημα. Δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει κανένα να κινηθεί προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Και αυτό το ζουν και οι Άγγλοι. Πολλοί έρχονται προς... Ε, πολλοί πάνε στην Αγγλία και πολλοί από τους Άγγλους φεύγουν. Γι' αυτό ρωτάμε καμιά φορά, γιατί θέλετε να πάρετε μέρος εσείς στο πρόγραμμα τους Βρετανούς. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να, να προσπαθήσουμε να το καταστήσουμε πιο ελκυστικό. Λοιπόν, κύριε Τόκιος, τον Ιανουάριο θα περιμένουμε την έκθεσή σας και μετά θα ψηφίσουμε. Ωραία. Πάμε στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης. Αναγνώριση και προώθηση των ε, διασυνοριακών δραστηριοτήτων ε, εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και επειδή αυτό το θέμα δεν έχει ιδιαίτερα ιδεολογικό περιεχόμενο, η πρώτη μας συνάντηση στην πρώτη συνάντηση άκουσα τις θέσεις και απόψεις των συναδέλφων ε, προκειμένου να καταρτήσω το κείμενο και να κανονίσω τη συνάντηση με τους κοιοδησηγητές. Δεν είμαστε και πολύ σε αυτή την αίθουσα, αλλά μπες ας προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε έχοντας κατά νου δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για εθελοντικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη επιτυχία και του Κοινοβουλίου μας. Θα ενθυμίσετε ότι όταν εξετάσαμε το Ευρωπαϊκό έτο Εθελοντισμού, η μεγάλη, η μεγάλη δυσκολία που είχαμε για πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, διότι δεν υπήρχαν οι νομικέ βάσει και ό,τι άλλο γνωρίζουμε και γνωρίζετε. Επανερχόμαστε λοιπόν στο ζήτημα των εθελοντικών δραστηριοτήτων που όπως γνωρίζετε έχει αποκτήσει διάσταση και στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Τώρα, η ανακοίνωση που έκανε η Κομισιόν είναι μια ανακοίνωση πολύ καλή, μια ανακοίνωση με την οποία συμφωνούμε και θέτει τις βάσεις ε, του όλου προβληματισμού. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε προκειμένου να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο ε, συνδέονται με κάποια ζητήματα που απ' όλα δεν υπάρχει ένα κοινό νομικό, μια κοινή νομική βάση ανάμεσα στα κράτη που αποτελούν ε, την, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα των διασυνοριακών εθνικών δραστηριοτήτων. Ε, μια άλλη πτυχή είναι η οικονομική πτυχή, διότι όπως τονίζει και η Κομισιόν, ε, ο εθελοντισμός ε, είναι δωρεάν, αλλά οι οργανώσεις, οι ενώσεις έχουν δαπάνες, οι οποίες αποτελούν και εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού που θα ξεπερνάει και τα σύνορα. Είχαμε την αρνητική εμπειρία της Ευρωπαϊκής ε, Εθελοντικής Υπηρεσίας σε ό,τι φορά το πρόγραμμα ε, νεολαία ενδράση η οικονομική στήριξη που δίνεται στους ε, εθελοντές είναι μια στήριξη η οποία προδικάζει μερικές φορές τη συμμετοχή σε κάποια μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί όπου οι δαπάνες είναι υψηλότερε και δεν επιτρέπουν στον εθελοντή να παίξει τον ρόλο του λόγω ακριβώς της έλλειψης οικονομικής στήριξης. Ένα κεντρικό θέμα είναι αυτό της αναγνώρισης των ε, των αρμοδιοτήτων ε, των... όταν ο εθελοντής ε, ασκεί το έργο του εκτός συνόρων, πώς θα μελετήσουν λοιπόν μία σειρά μέσων ε, που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του φαινόμενου τώρα. Το εμπόδιο, το φορολογικό, που είναι κάτι που συχνά διαφέρει από χώρα σε χώρα, δημιουργεί δυσκολίες για την ανάληψη κοινή ε, δράσης ε, και επίσης μια ανεπαρκής γνώση των στοιχείων και των εμπειριών των κρατών μελών. Από αυτή την άποψη λοιπόν ελπίζω ότι στο πέρας αυτού του τους εθελοντισμού, να μπορέσουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και να βρούμε κάποιες ε, αρχικές λύσεις αυτών των προβλημάτων που θα επιτρέψουν στον φάκελο αυτό να προχωρήσει και να δώσει πιο ουσιαστικές απαντήσεις. Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό της ελλειπούς γνώσης, δηλαδή πώς, τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να αποτανθούμε για τον, όταν θέλουμε να ασκήσουμε τον εθελοντισμό σε άλλα κράτη. Είτε πρόκειται για οργανώσεις είτε για μεμονωμένους εθελοντές, διότι υπάρχουν δυσκολίες το να γνωρίζουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να πετύχουν αυτό το στόχο τους. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό κατάλογο των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη τουλάχιστον σε επίπεδο εθελοντισμού ή τελίδα ή ένα γραφείο, μια υπηρεσία που να είναι κάπως πιο δομημένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπορεί να χορηγεί λοιπόν αυτές τις πληροφορίες και να επιτρέπει σε πρόσωπα και ενώσεις να δραστηριοποιούνται σε ζητήματα εθελονισμού. Και ε, αυτό που θα ήθελα να πω μετά αφού ακούσω τους συναδέλφους είναι να δραστηριοποιηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, διότι όπως σας είπα 100.000 είναι περίπου τα άτομα που ασχολούνται με τον εθελοντισμό στην Ευρώπη και εμείς ε, έχουμε ανάγκη να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω την δραστηριότητά του, διότι μέσω διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, να ε, πετύχουμε μια καλύτερη συνεργασία και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό μετά από τα όσα μα ε, διηγήθηκε σήμερα και η Επίτροπος Ρέντινγκ. Ευχαριστώ. Ποιο θέλει να κάνει παρατηρήσει, ο κύριος Ευχαριστώ. Αυτή είναι η δεύτερη έκθεση που έχει ως αντικείμενο την εθελοντική εργασία και την κάνετε πραγματικά πάρα πολύ επαγγελματικά, αλλά όπως είπατε υπάρχουν μεγάλα εμπόδια και αυτό έχει να κάνει με την αναγνώριση των προσόντων που έχουν οι εθελοντές. Οι εθελοντές που θέλουν να, είναι, να έχουν κινητικότητα, να ταξιδεύουν, να πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο και παρόλα αυτά να μπορούν να δουλέψουν ως εθελοντές. Σήμερα δουλεύουμε για, την, για το διαβατήριο των προσόντων για τους Ευρωπαίους, που θα αποτελεί μια εγγύηση. Ότι δηλαδή τα προσόντα τους αναγνωρίζονται και σε άλλα κράτη-μέλη και δεν ξέρω, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει έναν ε, τομέα που θα μπορούσε να καλύψει το, το διαβατήριο, δηλαδή να συμπεριλαμβάνεται στο διαβατήριο και η α, εθελοντική εργασία. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός τομέας δραστηριοτήτων για τους πολίτες μας. Ίσως λοιπόν να πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Μάρκους. Ε, πολλά από τα σημεία αναφέρθηκαν ήδη από εσά ό,τι αφορά τι αθλητικέ δραστηριότητε ε, και βεβαίω πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να βρούμε λύσει στα προβλήματα. Δύο πράγματα ήθελα εγώ να πω, τα οποία μου φαίνεται ότι είναι σημαντικά. Το ένα, το είδαμε σε σχέση και με, το, ε, με την έκθεση του Σαντιάγο για τον αθλητισμό, για τα προσόντα των εργαζομένων. Ε, σε κάποιες ε, περιπτώσεις δεν είναι σημαντικά, σε κάποια όμως σε κάποιες είναι, όπω όταν αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται μαζί με παιδιά, με νέους. Ε, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να έχουν και πρακτική εμπειρία, να έχουν γνώσεις πάνω στον αθλητισμό, εφόσον δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Το θέμα λοιπόν της χρηματοδότησης ή των των ε, προσόντων που έχουν ε, πρέπει να είναι ε, στοχοθετημένα τα προσόντα ανά τομέα. Επίσης, ένα άλλο που ήθελα να πω είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντών του χρόνου θα, του χρόνου θα είναι το έτος του, της του γυρα, της ε, γύρανσης ε, με ενέργεια. Ε, πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στο αυτό το σημείο να συμπεριλαμβάνεται. Αλλά, για παράδειγμα, τι γίνεται με τις δραστηριότητες εθελοντικές με, που είναι στο εξωτερικό, που προσφέρονται σε άλλες, ε, σε άλλες χώρες. Ε, μιλάμε για ανθρώπους που σε όλη τους τη ζωή εργάζονται εθελοντικά. Ε, βεβαίως ε, κοστίζουν πολύ λιγότερο γιατί έχουν προφανώς και καλές ε, συντάξεις αυτοί που δούλευαν στη ζωή τους και μπορούν να... να, να ζήσουν με αυτές, αλλά θα πρέπει να δούμε ίσως και την περίπτωση αυτή. Και αυτό το ερώτημα που είπε ο Μάρκος για το σημείο επαφή, Πού θα έχει κάποιο έναν συνομιλητή, πού μπορεί να πάει να βρει τέτοιε πληροφορίε ε, για να, θέλει, να μπορέσει να συμμετέχει αν θέλει. Νομίζω ότι ο θελοντισμός ξεπερνάει και την συνταξιοδότηση και την ηλικία συνταξιοδότηση. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν ε, και να δώσουν τα φώτα τους και, σε, και στους νέους ή να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να το σκεφτείτε έτσι λιγάκι και αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο θέμα του αθλητισμού θα πρέπει να διακρίνουμε τι είναι ο ε, εθελοντής και τι είναι ο τεχνικός. Ο τεχνικός έχει κάποιες ε, ικανότητες ε, συγκεκριμένες ε, που αφορούν τα συγκεκριμένα αθλήματα κλπ. Θα ήθελα επίσης στην έκθεση να, να συμπεριληφθούν και κάποια θέμα ασφάλειας, μια ασφάλισης των εθελοντών, διότι μπορεί να προκύψει, προκύψουν ευθύνες σε κάποιες δραστηριότητε που ενέχουν κινδύνους θα πρέπει λοιπόν να είναι ασφαλισμένοι. Τι, τι συμβαίνει αν ε, πέσουν ε, θύματα ατυχημάτων κλπ. Λοιπόν, σε αυτό το καθεστώς ε, του εθελοντισμού θα πρέπει να προβλέπεται και ένα είδος ασφάλισης που θα επιτρέπει να ασκήσει το όλο έργο του με κάποιες εγγύσεις ο Μία ιδέα της πέτρας θα ήθελα να σχολιάσω για το πώς μπορούμε να, προχωρη... να προωθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν όρεξη να προσφέρουν και πώς μπορούμε να τους δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες ε, για, τα, για κάτι για τη Γερμανία, ας πούμε, θα ήθελα να πω. Αν κάποιος ε, ε, προσφέρει κάτι για τους ε, μαθητές γυμνασίων, μπορεί μέσω επισκέψεων ή ταξιδιών να το προωθήσει, ας πούμε, να κάνει κονσέρτα ή για εκδηλώσεις σε βιβλιοθήκες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι καλό με τη βοήθεια της Κομισιόν να χρησιμοποιήσουμε τα δίκτυα που ήδη υπάρχουν και στα οποία μπορούμε να βασιστούμε και οι μη κυβερνητικέ είναι σημαντικέ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και να δούμε πού μπορούμε να βρούμε αυτού του ανθρώπου που θέλουμε να βρούμε και να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερες, ε, ε, περισσότερη δικτύωση από ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι στην προηγούμενη έκθεση είχα ζητήσει να μιλήσουμε και για το senior service και αυτό ακριβώς ε, λέμε, δηλαδή εθελοντική ε, εργασία των ηλικιωμένων. Ε, κάπου είδα σε μια ιστοσελίδα κάτι τέτοιο. Μπορεί να μην υπάρχει επαρκώ η προσφορά εθελοντική εργασία από ηλικιωμένου, αλλά νομίζω ότι κάπου υπάρχει. σω η Κομισιόν θα μπορούσε να μα πει κάτι από αυτού. Madame Sophie Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω σε κάποια από αυτά που ακούστηκαν σήμερα το απόγευμα. Όπως το υπογράμμισε και ο εισηγητής, το, η ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί πολιτική επιτυχία για την εθελοντική δράση, δεδομένου ότι για πρώτη φορά ενέκρινε ένα πολιτικό έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά αποκλειστικά την εθελοντική δράση. Όπως ε, γνωρίζετε, και εσείς θεωρούμε ότι είναι πράγματι πολιτική επιτυχία. Επίσης με ρώτησαν τα αποτελέσματα, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς, αυτού του έτους. Στο τέλος του 2012 θα, θα υπάρξει έκθεση που θα παρουσιάζει λεπτομερώς τα αποτελέσματα του έτους αυτού πέρα από την ανάλυση που λάβατε, από την ανακοίνωση που λάβατε, με συγχωρείτε και που αναλύεται τώρα. Τώρα όσον αφορά την αναγνώριση των αρμοδιοτήτων των, ε, και των δεξιοτήτων των ε, θελοντών υπάρχει αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη ένα ε, διαβατήριο που επιτρέπει να παραδιατηρηθεί το ίχνος των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Θα είναι το Aeropass ε, που θα μπορεί να το διατηρεί κανείς και να, να αποδεικνύει όλα αυτά. Όσον αφορά το θέμα της εθελοντικής εργασίας που προσφέρουν οι ηλικιωμένοι, υπάρχει ένα σκέλος του Grundwich που αφορά την ε, εθελοντική προσφορά των ε, ηλικιωμένων και φυσικά οι συνάδελφοι που θα αναλάβουν το 2012 για την ενεργό ε, γύρανση θα έχουν σημαντικό έργο να κάνουν στον τομέα αυτό της εθελοντικής προσφοράς των ηλικιωμένων που οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στους ε, νέους. Αυτά όσον αφορά το έτος 2012. Μετά αναφερθήκατε στο πώς θα ενημερωθούν οι πιθανοί θελοντές. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα έργα στα πλαίσια αυτού του έτους πολλές ενώσεις μεταξύ των οποίων η συμμαχία του 2011 δημιούργησε ένα σύστημα για να συσχετίσει τις προσφορές και τη ζήτηση. Και άλλοι το έχουν κάνει. Το Βέλγιο ας πούμε. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια αυτού του ευρωπαϊκού έτους. Ε, θα κλείσω στο σημείο αυτό, εκτός και αν έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Ευχαριστούμε προς το παρόν. Δεν ε, θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Οπότε θα συζητηθεί η έκθεσή σας ε, τον επόμενο Φεβρουάριο. Εντάξει. Εντάξει. Οπότε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν ε, σήμερα εδώ, όσοι ήσασταν εδώ. Είχαμε πολύ καλή εκπροσώπηση. Πάντα στο τέλος του χρόνου πρέπει να το λέω αυτό. Ήσασταν πάρα πολύ επιμελής. Το ξέρω γιατί ήμουν και εγώ στη θέση του κυρίου Σκουρία. Ευχαριστώ τον κύριο Σκουρία που ήταν τόσο καλός συντονιστής. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που ήταν παρόντες και οι πράσινοι προσωπήθηκαν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία όλους σας αυτή τη χρονιά. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να μην χωριστούμε για τα προγράμματα που πρέπει να προωθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δίκαιοι και ε, θα πρέπει και οι συντονιστές να προσπαθήσουν ώστε να μην πάμε να ικανοποιηθούμε και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στον επόμενο χρόνο. Καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα και καλή σας χρονιά. Σας ευχαριστώ όλους. So, Και τώρα συντονιστές.